favore prendiamo posizione. Καθίστε παρακαλώ. Benvenuti a tutti, cari όλοι, αγαπητοί εθνικοί βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη δεύτερη διακοινοβουλευτική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι πρώτη φορά στα 50 χρόνια ιστορίας της γεωργικής πολιτικής που οι βουλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην χάραξη του μέλλοντος της συγκεκριμένης πολιτικής. Το Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι συνομοθέτης στον τομέα της γεωργίας ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε μεγαλύτερες ευθύνες και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτό αυτή εδώ είναι η δεύτερη συνάντηση που είναι αφιερωμένη στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής που διοργανώνεται εντός ενός έτους. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συγκρίνουμε τις ιδέες μας, τις εμπειρίες μας για μια ευρωπαϊκή γεωργία πιο σύγχρονη. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση και στη νομιμοποίηση τη δημοκρατική της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εθνικούς βουλευτές τις πολυάριθμες συμβολές που έχετε στείλει στην Επιτροπή μας. Να θυμίσω ότι λάβαμε για αυτήν τη συνάντηση γραπτές συμβολές και γνωμοδοτήσεις από σχεδόν όλα τα εθνικά νομοθετικά σώματα. Επιπλέον μπορείτε να βρείτε ανάμεσα στα κείμενα το φυλάδιο της κατάστασης προόδου στα Εθνικά Κοινοβούλια για την κοινή γεωργική πολιτική και τη μεταρρύθμισή της. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινή γεωργική πολιτική αντιμετωπίζει προκλήσεις άνευ προηγουμένου σήμερα που επηρεάζουν την ζωή όλων μας. Ασφάλεια ανεφοδιασμού σε τρόφιμα έχει επανέλθει στην ατζέντα μας, στις προτεραιότητές μας. Λόγω της πλητικότητας των τιμών, την επιτάχυνση των κλιματικών αλλαγών, την αύξηση των πληθυσμών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι πριν τα παραγωγικά μας επίπεδα και την επάρκεια αυτών. Από την άλλη πλευρά, η πίεση στους φυσικούς μας πόρους ποτέ δεν ήταν τόσο έντονη. Οπότε προκύπτει ανάγκη μιας κοινή γεωργικής πολιτικής πιο πράσινης και πιο βιώσιμης. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε και το στόχο της παραγωγής υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αυξηθεί η στήριξη στην ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε η ανάπτυξη αυτή να είναι ισορροπημένη για όλες τις επικράτειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος οι Ευρωπαίοι Γεωργοί θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν κανόνες απλούς και όχι γραφειοκρατικούς με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις μεγάλες εξαγωγικές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική πιο ευέλικτη, πιο απλή στην εφαρμογή της και που θα λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία. Εύχομαι αγαπητοί συνάδελφοι πως η σημερινή συζήτηση θα είναι χρήσιμη. Θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην ανέβρεση λύσεων στα κοινά μας ερωτήματα, δηλαδή στις, μεγάλες, στις νέες μεγάλες προκλήσεις. Όπω ήδη γνωρίζετε, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει τι εργασίε του για αυτή τη μεταρρύθμιση τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ιούλιο του 2010 υιοθετήθηκε η πρώτη έκθεση για το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική μετά από το 2013 και εκεί εντοπίστηκαν οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου εν ώψη τη μελλοντική μεταρρύθμιση. Δηλαδή αυτό που εμεί αποκαλούμε έκθεση George Lyon, τον οποίο χαιρετώ. Ε, τον Ιούνιο του 2011 υιοθετήθηκε δεύτερη έκθεση ως επίσημη απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου 2010 για την κοινή γεωρική πολιτική. Έκθεση που φέρει το όνομα του Άλμπερ Ντες που είναι και εκείνος εδώ και τον χαιρετίζω. Στη συνέχεια η Κομισιόν δημοσίευσε τις νομοθετικές της προτάσεις επί της μεταρρύθμισης τον Οκτώβριο του 2011 και το Ευρωκοινοβούλιο όρισε τους εισηγητές του για κάθε τομέα. Μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με στόχο να συζητηθεί η πρόταση της Κομισιόν συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας ακρόσης με τον Επίτροπο Τσόλος, μια δημόσια συζήτηση με τους Υπουργούς Γεωργίας των 27 κρατών μελών, μια ακρόαση με ΜΚΟ, ε, και με ενδιαφερόμενους φορείς, μια διάσκεψη με εμπειρογνώμονες και καθηγητές και διάφορα σεμινάρια με, όπου μελετήθηκαν διάφορες πτυχές μεταρρύθμισης. Και τέλος, η σημερινή συνάντηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Την περασμένη εβδομάδα οι συγητές του Κοινοβουλίου για τις τέσσερις βασικές νομοθετικές προτάσεις ε, παρουσίασαν δημόσια τα σχέδια ε, προτάσεών τους ε, για την Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης. Λουίς Κάπουλα Σάντος για την ανάπτυξη Συπέθρου, ο Μισελ Νταντέν για την κοινή οργάνωση των αγορών, στα αριστερά μου κάθονται και οι δύο, και ο Τζοβάνι Λαβία για την χρηματοδότηση, έλεγχο και απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής που κάθεται δεξιά μου. Έχετε αντίτυπα αυτών των εκθέσεων στους φακέλους σας. Είναι εκθέσεις σημαντικές όπως μπορείτε να δείτε και ογκώδεις ε, και προβλέπουν εκατοντάδες τροπολογίες για αλλαγή, για διορθώσεις, για τροποποιήσεις της πρότασης της Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε, η παρουσίαση αυτών των εκθέσεων προκάλεσε μια πολύ ζωντανή συζήτηση στην Επιτροπή μας και στα κράτη-μέλη και μάλιστα περιμένουμε πολλές τροπολογίες ε, εν ώψη της συμπλήρωσης των εκθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και επιπλέον όχι μόνο η Επιτροπή Γεωργίας αλλά και διάφορες άλλες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ε, εμπλέκονται όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Περιφερειακών, ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Επιτροπή Ανάπτυξης, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η Επιτροπή Προϋπολογισμού όλες οι ιδέες που είναι επιτάπητος θα συζητηθούν πριν να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο την θέση του. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξή, ότι ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε η Επιτροπή Γεωργία, τη οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, θα μπορέσουν να υιοθετήσουν την, την τελική του έκθεση πριν από τη συμφωνία για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που θα διέπει την περίοδο 2014-2020. Εμείς αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικέ λύσει όσο γίνεται πιο σύντομα και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία το αργότερο τον φθινόπωρο, αλλά δεν θα προχωρήσουμε σε τελική ψηφοφορία μέχρι ότου να έχουμε τα στοιχεία για τον μελλοντικό προπολογισμό. Αγαπητοί λοιπόν συμμετέχοντες σε αυτή την ε, συνεδρίαση, δεδομένης τη κατάσταση πρόοδου τη μεταρρυθμίση, χρειάζεται να προτείνουμε πρακτικέ ιδέε που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το νομοθετικό πακέτο που πρότεινε η Κομισιόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα ζητήματα και γι' αυτό προτείνω να εστιάσετε τις παρεμβάσεις σας στα επιχειρήματα που αναφέρονται στο σημείωμα προσανατολισμού που έχετε λάβει και να εστιαστείτε δηλαδή περισσότερο στην κατανομή των άμεσων πληρωμών, σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και σε εσωτερική σύγκληση ανάμεσα στις περιφέρειες, κάπινγκ, δικαιούχοι των άμεσων πληρωμών, δηλαδή ο ενεργός γεωργός, οι νέοι γεωργοί, οι μικροί γεωργοί, πρασίνισμα στις άμεσες πληρωμές, υποχρεώσεις ε, και πρακτική εφαρμογή, όροι, ε, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσα για τη διαχείριση του κινδύνου, μέσα για την ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών, οι συμβατικές ε, εξουσίες των γεωργών και χρηματοδότηση της ε, αγροδιατροφικής, του αγροδιατροφικού τομέα. Επίσης, μέσα όπως οι ποσοστώσεις, ποσοστώσεις ζάχαρης, γάλακτος ή δικαιώματα φύτευσης για τα κλίματα. Ε, ελπίζω λοιπόν και εύχομαι αυτή η συνάντηση να προσδώσει ε, πρακτικές λύσεις για τους γεωργούς μας και τελικά να ωφελήσει το σύνολο των Ευρωπαίων γεωργών και των Ευρωπαίων πολιτών κατά συνέπεια. Όπως γνωρίζετε η απλοποίηση είναι ένα θέμα κλειδί και για να επιτύχουμε αυτό το στόχο ενδιαφερθήκαμε, θα, θέλουμε μάλλον να ακούσουμε τις διάφορες και καλύτερες πρακτικές που ε, εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Τέλος, συνάδελφοι, κάποιες ευκρινήσεις διαδικαστικού τύπου. Όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα βρουν στα έδρανά τους ένα έντυπο εγγραφής για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Σας καλώ λοιπόν να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να το δώσετε στους κλητήρες όσο γίνεται πιο σύντομα στους, επιτροπέ, στους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας να διευκρινίσω ότι και εκείνοι θέλουν, θα πρέπει μάλλον να συμπληρώσουν το εν λόγω έντυπο για να πάρουν το λόγο. Έχουμε εδώ παρόντες 47 ε, βουλευτές από 40, από σώματα και που αντιπροσωπεύουν 22 κράτη-μέλη. Ίσως να μην μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους το λόγο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε τουλάχιστον να γίνει μία παρέμβαση ανά σώμα οι παρεμβάσεις θα κατανεμηθούν ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Δύο παρεμβάσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μία παρέμβαση από το Ευρωκοινοβούλιο. Αν δεν αρκέσει ο χρόνος, προτεραιότητα θα δοθεί στους φιλοξενούμενούς μας. Για να γίνει αυτό δυνατό, θα σας παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά αναπαρέμβαση. Θα σας δίνω ενδείξεις, κατά τη, θα σας πω μάλλον πώς θα εκτεληθεί η κατά τη διάρκεια της. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον ε, πρόεδρο Ρενέ Κρίστενσεν, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Τροφίμων Γεωργίας και Αλληλείας του Δανέζικου Κοινοβουλίου, της Προεδρίας δηλαδή. Ευχαριστούμε κύριε Κρίστενσεν και σας δίνω Ευχαρίστω το λόγο για να ξεκινήσετε, να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών της συνόδου αυτής. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω πρώτα απ' όλα ποιος είμαι, ποιον εκπροσωπώ, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος της δανέζικης κυβέρνησης. Είμαι από το Λαϊκό Δανέζικο Κόμμα και είμαι στην αντιπολίτευση στη Δανία. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν ε, με το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, με το οποίο συμφωνούμε με την Προεδρία μας. Για τα περισσότερα σημεία υπάρχει συνένεση. Οπότε τι ήρθα να κάνω εδώ θα μου πείτε. Ε, λοιπόν, μία από τις προκλήσεις που θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασίας είναι ότι στο μέλλον, το είπε και ο Πρόεδρος, θα έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτές, στη ζήτηση δηλαδή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις μεγάλες αγορές και το μεγάλο δυναμικό που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τι ακριβώς θα γίνει. Πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή, ναι, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τη φύση και το περιβάλλον. Είναι αυτοί δύο αντιφατικοί ίσως στόχοι, λένε μερικοί. Δεν συμφωνώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ καλές δυνατότητες για να συνεισφέρουμε θετικά στην πρόταση αυτή, αλλά έχουμε και προκλήσεις μπροστά μας, όπως επίσης και ευκαιρίες. Γι' αυτό και είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν επιδοτήσεις οι αγρότες υπέρ του περιβάλλοντος και της οικολογικής παραγωγής. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και να προχωρήσουμε με καινοτόμε ιδέες. Χρειάζεται και τεχνικός εξοπλισμός βέβαια για να είναι πιο αποτελεσματική η γεωργία μας και να τα αποκρίνεται καλύτερα στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Το θέμα της τεχνολογίας πρέπει να συμπεριληφθεί στη συζήτηση αυτή. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστική γεωργία, η γεωργία μας να είναι βιώσιμη. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες ενισχύσεις όπως και τώρα στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι αγρότες πρέπει να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό ζητούν. Πρέπει να επικεντρωθούν στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας σε ολόκληρο τον ε, αγροτροφικό τομέα. Αυτή είναι μια πρόταση που είναι αλήθεια ότι την βλέπουμε και στις αρχές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη στηρίζω όλος ιδιαίτερος. Τώρα για τις άλλες προτάσεις που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, είναι το θέμα του 7% αγροτικής επιφάνειας που πρέπει να αφιερώνεται στο περιβάλλον ή στα βοσκοτόπια. Νομίζω ότι πρέπει να προβλέψουμε περισσότερη, περισσότερες ενισχύσεις και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό τοπίο. Η Προεδρία πρότεινε κάποια πράγματα για το πρασίνισμα, για την διάσταση της οικολογικότερης παραγωγής και οι περισσότεροι αγρότες συμφωνούν. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την απέτηση πρασινίσματος της παραγωγής, αλλά πρέπει να βασιζόμαστε και στους δύο πυλώνες και να μπορούν να έχουν εθνικές πιστοποίησεις οι ε, αγρότες. Και μερικές φορές σε εθνικό επίπεδο οι προδιαγραφές είναι πιο αυστηρές. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παραμείνει. Οι αγρότες πρέπει να μπορούν να διαλέξουν. Να διαλέξουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώνονται για να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους. Η σημερινή πρόταση της Κομισιόν λέει ότι πρέπει 7% να αφιερώνεται κυρίως στο περιβάλλον. Η Προεδρία λοιπόν έκανε μια πρόταση η οποία μας επιτρέπει να κατέβουμε στο 3,5% εφόσον το κράτος μέλος προβλέπει επιπλέον μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος, προγραμματικά μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος που να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη δηλαδή πρέπει να βρούνε τις ε, ζώνες που προτιμούν έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και όχι να μιλάμε για αυτό το 7% που θα είναι ένα μικρό κομματάκι σε κάθε ε, αγροτική εκμετάλλευση. Νομίζω ότι έχει να κερδίσει η Γεωργία από την δικιά μας την πρόταση. Τώρα για τους ενεργούς αγρότες. Αυτός που κρατάει την ε, εκμετάλλευση πρέπει να μπορεί να αποφεληθεί και από τις ενισχύσεις. Δεν πρέπει να αποκλείουμε κάποιους. Βλέπετε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις ενισχύσεις για να φτιάξουμε γήπεδα γκολφ ή για άλλους λόγους που δεν έχουν καμιά σχέση με την γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Η Επιτροπή θεώρησε ότι το πρασίνισμα θα οδηγούσε σε μία μείωση κατά 3% στο εισόδημα των αγροτών. Άρα έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Γεωργία γενικότερα. Όσον αφορά τώρα την παρέμβαση για μια κακή χρονιά, η Επιτροπή θα μπορούσε να βοηθήσει με την αποθήκευση. Αποτελεί δίκτυ ασφάλειας αυτό. Είναι τώρα η καλύτερη λύση, πρέπει μια τέτοια λύση να την κρατάμε για πολύ καιρό. Έχουμε προσφύγει σε τέτοια λύση κατά το παρελθόν, αλλά το θέμα της επαναγοράς δεν ξέρουμε αν θα αποδειχθεί αναγκαίο και στο μέλλον. Πρέπει να μπορούμε πρώτα να ανταποκριθούμε στη ζήτηση που υπάρχει για τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Άρα χρειαζόμαστε την καινοτομία και πρέπει να είμαστε σε θέση να παλέψουμε στις αγορές. Πιστεύω ότι η Δανέζοι και η Γεωργοί είναι φιλελεύθεροι και πιστεύω ότι το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συνεχίσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Γεωργία να προχωρήσει θετικά. Πιστεύω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Γεωργία πρέπει να δει πώς θα αυξήσει την παραγωγή, λαμβάνοντας όμως υπόψη και το περιβάλλον και τη φύση και το κλίμα. Στην Κοπεχάγη πρόσφατα σε μια κοινοβουλευτική συνάντηση που είχαμε, είπαμε ότι αν πίνανε ένα ποτήρι γάλα ε, οι Κινέζοι, αυτό θα αποτελούσε μια τεράστια αγορά για μας. Άρα πρέπει να δούμε πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μειώσουμε τον ε, προϋπολογισμό ε, που πάει στη Γεωργία, αλλά να βελτιώσουμε την έρευνα για να βελτιώσουμε την παραγωγή και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και το κλίμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων για το περιβάλλον και την οικολογία. Τέλος, πολύ σημαντικό, πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες που να είναι στραμμένες προς την οικολογία. Η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί. Όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να βελτιώσουν το πρασίνισμα της παραγωγής με άμεσες ενισχύσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Είμαι ο πρώτο που παίρνω το λόγο εδώ σήμερα και βλέπω πολλά πρόσωπα στην αίθουσα που γνωρίζω ήδη και που είδα και στη διακοινωνευτική συνάντηση που είχαμε στην Κοπεχάγη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε μια καρποφόρα συζήτηση και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε εκεί, παρόλο που η μερίσια διάταξη εδώ σήμερα είναι κάπως διαφορετική. Ελπίζω όμως ότι θα προχωρήσουμε για να ανταποκριθούμε στους στόχους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία σήμερα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε Κρίστενσεν. Και τώρα πριν να δώσω το λόγο στους ε, τρεις εισηγητές μας ε, με τη σειρά Κάπουλα, Σάντος, Νταντέν και Τζοβάνι Λαβία ήθελα επίσης να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους 24 ε, φοιτητές της νήσου Λαπάλμα που ήρθαν για να συναντήσουν την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, Λουίς, έχεις το λόγο για να παρουσιάσεις την έκθεσή σου. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντα όλους τους συναδέλφους. Είναι μεγάλη χαρά να μπορούμε να τους υποδεχόμαστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι αυτή η σημερινή μας συνεδρίαση θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας και ότι θα μπορέσουμε να έχω, βρούμε μια συνένεση όσο γίνεται ευρύτερη για την ευρωπαϊκή, μελλοντική ευρωπαϊκή γεωργία. Οι δύο εκθέσεις, ε, τις οποίες ε, ανέλαβα να υλοποιήσω και τις οποίες γνωρίζετε, δεν αντικατοπτρίζουν φυσικά αυστηρά την προσωπική μου γνώμη. Δούλεψα εδώ και 6-7 μήνες, έχω μιλήσει με σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις, με πολλές περιφερειακές κυβερνήσεις, με σχεδόν όλες τις ομοσπονδίες και συνεταιρισμούς του γεωργικούς, με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και προσπάθησα να φτιάξω ένα, ε, να βρω μια ισορροπία ώστε να βρεθεί συνένεση. Φυσικά οι συμβιβασμοί γενικά ε, δυσαρεστούν όλους, αλλά η μέθοδος ε, κοινοτική δεν επιτρέπει άλλο δρόμο. Γι' αυτό θα ήθελα να ερμηνεύσετε τις προτάσεις μου ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε, να καταφέρουμε στην μελλοντική Ευρώπη να συνδυάσουμε την παραγωγικότητα με την βιωσιμότητα και να διατηρήσουμε την ε, ζωντάνια, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική στις ε, περιοχές της υπαίθρου. Θα ήθελα η πρότασή μου να είναι πιο δίκαιη και πιο ισότιμη από την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την ανακατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη μέση βοήθεια ανά εκτάριο ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Μια διαφορά που φτάνει πάνω από το 50% ε, ε, ε, από μέσες αξίες πάνω από το 60% υπάρχουν κράτη-μέλη που, που ισχύει και υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι 50% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η αξία αυτή. Εγώ προσπάθησα λοιπόν έτσι ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση των κρατών που βρίσκονται στη χειρότερη θέση ε, στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή οι βαλτικές χώρες, έτσι ώστε στην πρότασή μου ορισμένες από αυτές διπλασιάζουν, διπλασιάζουν τα ποσά που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ε, και ακόμα και έτσι βρίσκονται 35% κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο Πράγμα το οποίο είναι <laughs> άδικο, κατά τη γνώμη μου. Ε, επίσης προσπάθησα να ε, εντάξω περισσότερο ρεαλισμό και δικαιοσύνη μέσα σε κάθε κράτο μέλος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αργεί πολύ με τις προτάσεις της όσον αφορά την ανακατανομή εντό των κρατών μελών των ιδίων είναι πολύ ταχεία. Γι' αυτό προσπάθησα να υπάρξει πιο γρήγορα σύγκληση μέσα στα ίδια τα κρατημέλη και να υπάρχουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν εντός των ίδιων των κρατών μελών και εντός των περιφερειών να αποφύγουν ορισμένοι τομείς να συναντήσουν μεγάλη πτώση των, της απόδοσης, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις δραστηριότητες στα συγκεκριμένες περιφέρειες ή στα κρατημέλη. Απ' την άλλη πλευρά προσπάθησα στο πρώτο πυλώνας και, ο, και η κοινή γεωργική πολιτική να γίνουν πιο πράγματα πράσινα. Εμείς ε, έχουμε αυτό το καθήκον απέναντι στην κοινωνία. Οι γεωργοί πρέπει να στηριχθούν από δημόσια κονδύλια, πρέπει να ανταμυφθούν, αλλά και θα πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν μια υπηρεσία στους πολίτες μέσω της παροχή ε, δημοσίων αγαθών που μπορούν να παράγουν ε, και γι' αυτό αυτή η κοινή γεωργική πολιτική θέλουμε να είναι καταπράσινη καταπράσινη όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και πιο απλή. Όλοι μας μιλάμε πολύ για απλοποίηση, αλλά όταν πρόκειται Μάλλον τη στιγμή που θέλουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένα μέτρα απλοποίηση, συνήθω δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ προσπάθησα λοιπόν να εισάγω εδώ πραγματικά μέτρα απλοποίηση, όπω θα σα το δείξω κιόλα έτσι εν συντομία. Θα ήθελα λοιπόν, συντομία να σας πω, ότι σε σχέση με το θέμα του ενεργού αγρότη έχω εισάγει μια μεγάλη ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν αλλά πάντοτε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γεωργός είναι αυτός που ασκεί μια γεωργική δραστηριότητα, σημαντική. Σε σχέση με το πρασίνισμα Διατήρησα την αρχιτεκτονική της Κομισιόν κατά βάση, αλλά ε, έχω εισάγει κάποιες νέες πτυχές. Καταρχήν, εισαγωγή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του δεύτερου πυλώνα ως προϋπόθεση πρόσβασης στο πρασίνισμα. Επίσης, όρες όπως η Κομισιόν είχε προτείνει με την, ε, για την βιολογική γεωργία. Από την άλλη πλευρά, ε, εισάγουμε ένα σύστημα αντιστοιχίας, δηλαδή δυνατότητα των κρατών μελών επί τη βάση ενός κοινοτικού κανονισμού να μπορούν να πιστοποιούν οικολογικά τις παραγωγές αυτές και με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθώ στους συναδέλφους που ήθελαν να υπάρχει ένα μενού, ένας κατάλογος μέτρων πιο ευρύς που θα ήταν όμως αδύνατον να συζητήσουμε τα μέτρα αυτά ένα προς ένα γιατί αν ε, λάβουμε υπόψη την ε, αντιπαράθεση που προκάλεσαν τα τρία μέτρα μόλις που πρότεινε η Κομισιόν, φανταστείτε τι θα γινόταν αν αντί για τρία μόλις μέτρα είχαμε 10-15 μέτρα. Γι' αυτό και ε, θέλω να εισάγω ένα σύστημα αντιστοιχίας, δηλαδή τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου και τη δυνατότητα των κρατών μελών να ορίζουν και να καθορίζουν τον τρόπο οικολογικής πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου θα αναγνωρίζεται ότι τηρούν τις απαιτήσεις του greening. Έπειτα, δέχομαι και μέτρα της Κομισιόν, ας πούμε, για, συμπληρώνω μάλλον τα μέτρα της Κομισιόν για τις οικολογικές ε, καλλιέργειες να εφαρμόζονται αυτά τα, αυτοί οι όροι στις εκμεταλλεύσεις άνω των 20 εκταρίων, έτσι ώστε να καλύπτεται το 80% των γεωργικών ε, επιφανειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 80% το υπογραμμίζω και το ξαναλέω. 80% των γεωργικών επιφανειών να υποβληθούν στα μέτρα πρασινίσματος. Αλλά και αυτές έτσι φτάνουμε στο 80% των γεωργών και είναι δυνατόν να απελευθερωθούν έτσι από το γραφειοκρατικό φόρτο και το σύστημα ελέγχου ένας μεγάλος αριθμός γεωργών των των οποίων η συμβολή για την ε, οικολογία θα ήταν μικρή και ενώ από πλευράς γραφειοκρατικής θα ήταν τεράστιος ο φόρτος και θα υπήρχαν μεγάλες επιπλοκές. Έπειτα προτείνω να απλοποιηθεί το σύστημα των ε, ζωνών οικολογικού ενδιαφέροντας, δίνοντας στους γεωργούς τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν αυτές τις ζώνες που δεν είναι παραγωγικές με ζώνες παραγωγής ε, συγκεκριμένων ε, φυτών που απορροφούν το άζωτο από το έδαφος. Αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία περιβαλλοντική και επιτρέπει να διατηρήσουν την παραγωγή τους ε, γες με μεγάλη παραγωγικότητα που διαφορετικά θα αποκλείονταν. Επίσης εισάγεται δυνατότητα πάντοτε επειδή ε, δύο ε, επειδή μπορούν να υπάρχουν ε, ζώνες μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος, να είναι τα ποσοστά μικρότερα. Για τους νέους γεωργούς επίσης εισάγουμε ένα σύστημα top-up που η Κομισιόν προτείνει να εφαρμόζεται για μια περιοχή ίση σε κάθε κράτος μέλος και όχι μεταβλητή σύμφωνη με, τη μέση, με το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε κάθε χώρα. Απλοποιώ το σύστημα και βελτιώνω το σύστημα των νέων γεωργών που το καθιστώ εθελοντικό, προαιρετικό έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται στις χώρες μέλη όπου το πρόβλημα επίγει και επίσης προτείνω έναν μηχανισμό ευελιξίας ανάμεσα στους δύο πυλώνες να είναι πιο εύκολο και πιο συνολικό για να μπορεί να γίνει να μπορούν να υπάρχουν μετακινήσεις από τον ένα πυλώνα στον άλλον κονδυλίων και να μπορούν να λαμβάνονται ευρύτερα μέτρα μέσω του δεύτερου πυλώνα. Και επειδή έχω ακόμα μόνο ένα λεπτό, να πω στο, στο, στην έκθεση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Κανονικά θα ήθελα άλλα δύο-τρία λεπτά, Πρόεδρε, αν και προσπαθώ να είμαι πολύ γρήγορος. Σε σχέση λοιπόν με την ανάπτυξη της υπαίθρου, αυτό που προτείνω είναι βασικά το εξή. Προτείνω το 30% του προπολογισμού να αφιερωθεί σε, ε, σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Δηλαδή μπαίνουν αυτά στο πρώτο πυλώνα του greening, αλλά είναι απαραίτητο στο δεύτερο πυλώνα να υπάρχουν κονδύλια κατάλληλα που να συνοδεύουν αυτό το μέτρο. Προτείνω επίσης να εγκαταστεί ευρύτερη στήριξη στους νέους γεωργού στο δεύτερο πυλώνα, εισάγοντα ε, μηχανισμούς που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη. Γιατί η πρόσβαση στη γη είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης των γενεών. Ε, γι' αυτό και με, εισάγω και ένα νέο μηχανισμό απόσυρση από τη δραστηριότητα. Οι γεωργοί πάνω των, άνω των 50 ετών να μεταφέρουν την ε, εκμετάλλευτή του σε ένα νέο ε, αγρότη, έτσι ώστε να τους, και μάλιστα σε αυτού να δίνεται ένα 50% του ποσού που αποδίδεται στην εγκατάσταση ενό νέου γεωργού. Επίσης προτείνω τη διευκόλυνση του επίμαχου θέματα του ορισμού των ε, ζωνών με φυσικού ορισμούς. Η Κομισιόν προτείνει κριτήρια βιοφυσικά. Ε, αυτό όμως θα οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις στο δικαστήριο. Εγώ λέω να σεβαστούμε αυτά τα κριτήρια, αλλά να αφήσουμε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κρατών μελών ε, δεν έχει δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να γνωρίζουμε ακριβώς τις συνέπειες μιας τέτοιας πρότασης που υπέβαλε η Κομισιόν. Στο δεύτερο πυλώνα ε, ε, προτείνω επίσης να καλυφθεί μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κενό γιατί η Κομισιόν δεν προτείνει ε, κατανομή. Η κλίδα της κατανομής να διατηρηθεί όπως ισχύει. Όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στη χειρότερη θέση στο δεύτερο πυλώνα είναι εκείνα τα οποία είναι στην καλύτερη θέση στον πρώτο πυλώνα. Οπότε, οποιοδήποτε μηχανισμός αφαιρούσε από τα κράτη-μέλη που είναι σε καλύτερη θέση στο δεύτερο πυλώνα, βαλτικέ χώρε, για παράδειγμα, τα χρήματα κάθε ολόκληρο του, προ... του προπολογισμού αυτών των χωρών δεν θα έφτανε για να διορθωθεί κάπως η κατάσταση στη Γαλλία, στη Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν, επειδή ο δεύτερος πυλώνας είναι μόλις το 25% του συνολικού κονδυλίου, πιστεύω πως η πιο δίκαιη λύση είναι να διατηρήσουμε την ε, κατανομή όπου κανένα κράτος μέλος να, μην δει, να μειώνει το προπολογισμό του σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Υπάρχουν ακόμα προτάσεις για τα δάση, για τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις στην ε, ε, βιομηχανία του τομέα, ευρύτερη κατανομή. Αυτές είναι συνοπτικά οι βασικές ε, προτάσεις. και ε, περιμένω τις δικές σας συμβολές και εναλλακτικέ λύσεις γιατί φυσικά αν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικέ λύσεις είμαι διαθέσιμος να τις δεχτώ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε, που είναι, ε, να επιτύχουμε τους στόχους μας περισσότερη απλοποίηση, περισσότερη δικαιοσύνη περισσότερη πράσινη κυνηγερική πολιτική πιο δίκαιη και ισότιμη για τους γεωργούς και για τα κρατημέλη Σας ευχαριστώ σε ευχαριστούμε Λουίς και ευχαριστούμε για την ε, προσπάθεια που έκανα σας να τα πεις πιο συναπτικά γιατί οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το, ίσως το πιο ε, λεπτό θέμα, τα πιο λεπτά θέματα μέσα στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης. Να χαιρετήσω και τους εκπροσώπους ε, της χώρας μου, γιατί ανάμεσα στους 47 ε, εθνικούς βουλευτές είναι παρόν ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Ιταλικής Γερουσίας κ. Κάπα και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τους χαιρετίζω και τους δύο. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Μισελ Νταντάν, στον οποίο θα ζητήσω επίσης να είναι σύντομος γιατί προ... αν λάβουμε υπόψη τις 400 τόσες αλλαγές που προτείνει στην έκθεσή του, δεν θα είναι εύκολο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας ε, καλωσορίσω και εγώ και θα σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που δεχθήκατε την ε, πρόσκλησή μας. Πρέπει να στήσω συγγνώμη εκ των Γάλλων ε, συναδέλφων, οι οποίοι έχουν βρεθεί παγιδευμένοι σε ένα τρένο λόγω κάποιου τυχήματος στη γραμμή Παρίσι-Βρυξέλλε και έτσι δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν ακόμη. Η κοινή οργάνωση των αγορών λοιπόν είναι μια έκθεση σημαντική διότι η οικονομική, η γεωργική δραστηριότητα παραμένει πάνω απ' όλα οικονομική. Στην τελευταία δεκαετία άλλαξε ριζικά ο κόσμος μας και οι γεωργικές μας παραγωγές πλήττονται από το φαινόμενο της πτυτικότητας των τιμών τόσο για τα ε, προϊόντα που προσφέρονται για πώληση αλλά και όσο για την επιβάρυνση στην οποία εφίσταται ε, μια γεωργική εκμετάλλευση. Και γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε για να ενδοθούμε από τις, από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία 20 χρόνια και ενδεχομένω να καταλήξουμε κάποια ανάλυση για την ε, ρύθμιση των αγορών. Εν του εξελισσόμενου αυτού κόσμου σας προτείνουμε με τα όσα μας πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, ιδέες που εξέθεσε, να εξασφαλίσουμε ένα μέσον αντιμετώπισης κρίση αυτό που ονομάζουμε δίκτυα ασφαλεία, για να επιτρέψουμε στο Γεωργό να εξασφαλίσει μια, έναν έλεγχο πλήρη διεξοδικό της ε, θέσης του στην αγορά και τις ε, λειτουργίες της αγοράς αυτής. Για να το καταφέρουμε όμως αυτό δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση της ίδιας της οργάνωσης. Χρειάζεται οι εξουσίες που έχουν χορηγηθεί στις ε, οργανώσεις να υλοποιηθούν ουσιαστικά και επίσης θα πρότεινα να ληφθεί υπόψη η σημαντική αλλαγή που σημειώνεται. Δηλαδή από την εποχή όπου οι τιμέ όπω ορίζονταν έδιναν κατευθύνσει σε αγορές και που προσπαθούσαμε να εμποδίσουμε τον Γεωργό από την ανάληψη μια πρωτοβουλία που θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτές τις τιμέ που, ε, και που τώρα έχει μετατραπεί σε, δεδομένη, σε μια αγορά δεδομένης ε, ελεύθερης εμπορικής συναλλαγή. Άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνε για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία και δι' Πρώτον, επειδή το δίκαιο του ανταγωνισμού στις χώρες μας αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τρόπους σκέψης και δράσεις πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους και οι οποίοι εν τέλει ε, από κοινού παρεμποδίζουν την ε, πρόσκοπτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, νέας αγοράς. Επίσης, άπαξ και γίνεται η αγορά και οι οργανώσει των παραγωγών, ο, ο κατά κανόνα τρόπο λειτουργία των αγορών αυτών, θα πρέπει να διευκρινιστούν και να διασαφινιστούν, να εξασφαλιστούν οι πρωτοβουλίε των οργανώσεων αυτών, των συμφωνιών μεταξύ παραγωγών και της αλυσίδας της ε, διοχέτευσης των ε, προϊόντων, έτσι ώστε να λειτουργεί καλά η αγορά. Η δουλειά αυτή βέβαια είναι μια δουλειά λεπτή, Πρέπει όμως να υπενθυμίσω ότι και στη συνθήκη της Ρώμης το 57 αλλά και στη συνθήκη της Λισαβόνας το άρθρο 42 προβλέπει ότι τα συμβαλόμενα μέρη προβλέπουν τη δυνατότητα της ε, θέσπισης ρυθμίσεων για το δικαίωμα του ανταγωνισμού κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και εγώ καλώ ε, τους ενδιαφερομένους να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της δυνατότητας. Ευχαριστώ πολύ Μισελ. Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη δική μου έκθεση προσπάθησα με κάθε τρόπο να ε, εστιάσω τις ε, αλλαγές προς την κατεύθυνση της απλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση προσπάθησα όσον αφορά τη διαχείριση και την, ε, τον έλεγχο της κοινή γεωργικής πολιτικής η απλοποίηση αυτή να είναι το βασικό στοιχείο. Γι' αυτό προσπάθησα να εστιάσω την προσοχή σε ορισμένες πτυχές. Καταρχήν αυτή που σχετίζεται με την παρουσία των ε, αιτήματων. Κάθε φορά υποχρεώνουμε τις ε, εκμεταλλεύσεις να υποβάλουν αιτήματα κάθε χρόνο χωρίς να έχει αλλάξει, ακόμα μάλλον και αν δεν έχει αλλάξει κάτι στη δομή των ε, εταιριών. Να γίνεται λοιπόν μια απλή επιβιβαίωση της ε, συνέχισης της ίδιας δικασίας με στόχο την απλοποίηση του φόρτου για κάθε επιχείρηση ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να παράγουν όλο και περισσότερο χαρτί. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η απλοποίηση του ελέγχου και η μείωση των ελέγχων έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι οι εκμεταλλεύσεις και κυρίως τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών να δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρότεινα ως αλλαγή σε σχέση με την αρχική διατύπωση της Κομισιόν, πρότεινα ο ελεκτικός μηχανισμός να λειτουργεί μέσω μιας εσωτερικής και εξωτερικής πιστοποίησης πιο συγκεκριμένης, ούτως ώστε να μειώνονται τα κόστη ελέγχου που επιβαρύνουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, επίσης, και σε σχέση με τις κυρώσεις Έχω κάνει μια σημαντική τροποποίηση. Θα ήθελα δηλαδή οι κυρώσεις να είναι αναλογικές. Είδαμε στο παρελθόν ότι σε σχέση με μικρά, πολύ μικρά σφάλματα των γεωργών, ορισμένες φορές οι κυρώσεις που επιβάλλονταν ήταν πραγματικά δυσανάλογες. Με άλλα λόγια, μικρά σφάλματα τυπικού χαρακτήρα πολλές φορές τιμωρούνταν με κυρώσεις που σήμαιναν όχι μόνο την απώλεια της ενίσχυσης, αλλά και πολυετή ε, ποινή. Άρα λοιπόν πέρα από την αναλογικότητα της κύρωσης πρότεινα να φτιαχτεί ένα σύστημα προειδοποίησης αφού είμαστε σε μια περίοδο που όλοι μιλάμε και ενδιαφερόμαστε όλο ένα και περισσότερο για το ποδόσφαιρο, ένα είδος κίτρινης κάρτας, σε μια προειδοποίηση δηλαδή προς τον Γιώργο ότι δεν πρέπει να συνεχίσει με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά λανθασμένη. Με το σύστημα λοιπόν της έγκαιρης προειδοποίησης θα μπορούμε να μειώσουμε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις τελικές ποινές κυρώσεις προς τους γεωργιούς και να γλιτώσουν αυτοί που εν αγνία διαπράττουν σφάλματα στην εφαρμογή των πολιτικών. Ένα άλλο θέμα είναι το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα σε αυτό το κοινοβούλιο έχει συζητηθεί επί μακρόν και μετά από μια μακρά διαβούλευση με τους συναδέλφους, αφού αντιμετωπίσαμε στο εσωτερικό, μάλλον ε, συζητήσαμε και στο εσωτερικό της Επιτροπής, τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κυρίως στην πρώτη φάση εφαρμογής, δηλαδή σε αυτή την φάση όπου αυτό το νέο μέσο πρασινίσματος της κοινή γεωργικής πολιτικής θα αρχίσει να ισχύει, δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει ποινή η οποία να ξεπερνά την ίδια την πληρωμή του κομματιού greening. Δηλαδή προτείνεται να υπάρχει κύρωση στην περίπτωση μη εφαρμογή του περασινίσματος. Έχω προβλέψει μέσα στην έκθεσή μου το, η κύρωση να έρχεται στο ποσοστό του, ενίσχυση για το greening. Και σε συνεργασία με τον ε, συνάδελφο Καπούλας ε, Σάντος έχουμε διευρύνει τις, τις κατηγορίες ε, των γεωργών που αυτομάτως θα μπορούν να χαίρουν αυτών των κονδυλίων, της ενίσχυσης για το greening. Ε, Στην ε, πρόταση της Κομισιόν μόνο μπορούσαν ε, οι, οι βιολογικές καλλιέργειες να πάρουν το greening αυτόματα. Από τη στιγμή δηλαδή που παίρνουν το δεύτερο πυλώνα θα παίρνουν και τον πρώτο πυλώνα. Ενώ εμείς προτείνουμε μια απλοποίηση για όλες τις χώρες και κυρίως για αυτές που έχουν εσωτερική δομή η οποία είναι συνδεδεμένη με το περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη Σιπέδρου. εκεί έχουμε ακόμα ένα θέμα το οποίο ήδη είχαμε ε, εισάγει στον κανονισμό ευθυγράμμωση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα την προηγούμενη δηλαδή νομοθεσία, που αφορά την αποδέσμευση σε εθνικό επίπεδο. Πολύ συχνά σε μεμονωμένε χώρε που έχουν ε, λειτουργικά προγράμματα για την ανάπτυξη Σιπέδρου σε περιφερειακό επίπεδο, έχουμε κάποιε περιφέρειες που μπορούν να δαπανίσουν και δαπανούν και άλλες οι οποίες είναι πιο αργές, έχουν δυσκολίες και πολύ συχνά χάνουν πόρους. Η πρόταση λοιπόν προβλέπει μια αντιστάθμιση, μια δυνατότητα αντιστάθμισης σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της μεμονωμένης χώρες να μπορούν να αποζημιωθούν με μεγαλύτερες δυνατότητες δαπάνες ορισμένων περιφερειών, ε, ορισμένες αδυναμίες ε, που αντιμετωπίζονται σε άλλες περιφέρειες. Άλλα θέματα είναι οι όροι, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ε, αρχικό ήταν, αφορούσε την εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα και για τα ζυζανιοκτώνα μέσα στην πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο της ε, συναπόφασης και δεν μπορεί απλώς να εισαχθεί μέσα στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής στο εσωτερικό της, του κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου και κατά συνέπεια στον οριζόντιο κανονισμό υπάρχει το θέμα της καινοτόμας τοπικής συνεργασίας. Νομίζω πως αυτό όμως είναι κατά των αρχών, αντίθετο με τις αρχές ε, της εφαρμογής του προγράμματος LEADER και ε, αντίθετο με τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ε, χρηματοδότησης. Ε, υπάρχει δηλαδή αντίφαση ανάμεσα στα όσα υπάρχουν στη διαθεσή μας και αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν το έχω τροποποιήσει, αλλά ανέκαθεν σε κάθε συζήτηση που έχουμε κάνει στην Επιτροπή Γεωργίας έχω θέσει επιτάπητο στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αν φτάσουμε σε κάποια συνεννόηση, πιστεύω πως η συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Τζοβάνι και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση. Όπως είπαμε από την αρχή θα δώσω το λόγο σε δύο εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και έναν της Επιτροπής Γεωργίας του Κοινοβουλίου. Ε, μέχρι ότου μας το επιτρέπει ο χρόνος, γιατί διαφορετικά θα δώσω την προτεραιότητα φυσικά στους φιλοξενούμενούς μας, στους καλεσμένους μας. Θα σας θυμίσω λοιπόν το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Κυπριακού ε, Κοινοβουλίου, Γαβρίλ Γιαννάκης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γιαννάκης πρέγω. Κύριος Γαβρίλ Γιαννάκης, παρακαλώ, πιέστε το. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι, επιτρέψτε μου πριν να τοποθετηθώ να συγχαρώ του συζητητέ για την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργία και Φυσικών Μπορών αντιμετωπίζει θετικά τι βασικέ αρχέ στι οποίε στηρίζονται οι προτάσει τη Επιτροπή, επισημένοντα ταυτόχρονα την ανάγκη για ευελιξία, απλοποίηση και μείωση του διοικητικού φόρτου. Τονίζει επίση την ανάγκη όπω οι αναλόγω προτάσει τη Επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τι ιδιαιτερότητε του κάθε κράτου μέλου. Σε ό,τι αφορά τι άμεσε ενισχύσει, η Επιτροπή χαιρετίζει την αλληλογοπρόταση, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε να αποφευθεί η μείωση του δημοσιονομικού φακέλου των μικρών κρατών που αντιμετωπίζουν διαθροτικά προβλήματα λόγω μεγέθους αλλά και απόστασης από τις αγορές ενώ παράλληλα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή όπως η Κύπρος. Παράλληλα, θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη όσον αφορά το πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών τόσο ω προ την επιλογή των επιμέρου μέτρων, όσο και για σκοπού απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογή. Καλωσορίζει την εισαγωγή του ειδικού σχεδίου για του μικροκαλλιεργητέ, των οποίων ο ρόλο είναι σημαντικό για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί δυνατότητα σε μικρά κράτη-μέλη τα οποία διαθέτουν μεγάλων αριθμό μικροκαλλιεργητών να παρέχουν μεγαλύτερο ποσοστό από το δημοσιονομικό του φάκελο για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Αναφορικά με την πρόταση για την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή συμφωνεί με του τρει βασικού στόχου και προτεραιότητε τη πρόταση τη Επιτροπή και θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και απλοποίησης αυτής, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Τονίζει ότι θα πρέπει να αποφευθούν οι επικαλύψει μεταξύ του πρασινίσματο των άμεσων πληρωμών και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματο αγροτική ανάπτυξη. Τέλο, χαιρετίζει τι πρότεινε που επιτρέπουν στην Επιτροπή να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για αντιμετώπιση μεγάλων διαταραχών στην αγορά με χρηματοδότηση από το Ταμείο Διαχείριση Κρίσεων. Τονίζει τη σημασία καθορισμού ξεκάθαρων κριτηρίων για την ενεργοποίηση των μέτρων αυτών ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να υποφεληθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας ε, της ε, Βουλής των Κοινοτήτων, Άννα Μάκιντος. Έχεις το λόγο, Άννα. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια στην Προεδρία της Δανίας, την απερχόμενη, αλλά και καλώς ήρθατε στην καινούρια Προεδρία της Κύπρου. Πολύ είναι το κοινό πεδίο μεταξύ των ε, επόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. όλός θα παρουσιαστούν και σήμερα εδώ. Μπορώ να συμφωνήσω με τους ηγητές ότι κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο απλή κοινή πολιτική με περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Οι ιδέες λοιπόν της Προεδρίας της Δανίας για την πιστοποίηση για μας γεννούν κάποιες ανησυχίες με την έννοια ότι μπορεί να ε, οδηγήσουν σε περισσότερη γραφειοκρατία ως εκ τούτου και θα καλέσω τους συναδέλφους να διαβάσουν το έγγραφο της Βουλής των Κοινοτήτων ε, όπου υπογραμμίζεται ότι ο κέριος στόχος μας είναι να περιοριστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή λέει, θα ορίζει τους γενικότερους στόχους και κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους σε συνεργασία με τους γεωργούς της θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο να ορίσει, προς την να ορίσει το, ε, τα πραγματικά πράσινα μέτρα που θα εισαγαγεί. Όπω είπε και ο κ. Καπούλα Για ένα από τα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω, που δεν είχα την ευκαιρία να αναφέρω στην ε, Κοπενχάγη, οι μεταφορέ από, το από τον πλώνα 1 στον πλώνα 2 ήδη προξενούν δυσκολίε και φέρνουν σε μειονεκτική θέση του γεώργου τη Βρετανία και πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Οποιασδήποτε συστήσει λοιπόν γίνουν και σήμερα και στου επόμενου 6 μήνε θα πρέπει να μην επισκέστον από το γεγονό ότι ακόμη δεν έχουν αποφασίσει οι υπουργοί στο Συμβούλιο για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πολύ βασικό είναι εμεί να διατηρήσουμε ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία μεταξύ μα. Σα ευχαριστώ κυρία Μάκιντο. Και τώρα η κυρία Κέστιγκερ, βουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ξαναπεράσουμε μετά στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρία Κέστιγκερ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ ρητά να αναφέρω ότι θεωρώ πολύ καλή την ευκαιρία που μας προσφέρεται σήμερα να συστήσουμε με τους συναδέλφους από τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι πολύ σημαντικό να συνέρχονται στην ίδια συνεδρίαση τα Εθνικά Κοινοβούλια Φενό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Φετέρου για να συζητήσουν κάθε μία από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και να δράξουν κάθε δυνατή ευκαιρία. Έτσι λοιπόν αυτή η κοινή συνεργασία, αυτή η κοινή διαμόρφωση της γεωργικής πολιτικής νομίζω μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον για μια πιο αποτελεσματική πολιτική. Πρέπει βεβαίω να διατεθούν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Κάθε πιθανή περικοπή που ενδεχομένως προτείνεται στη γεωργική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη πέθρου, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι ο κύριος ε, Καπούλα Σάντος αξίζει συγχαρητηρίων για τις προσπάθειές του και την επιτυχία του στον τομέα αυτών, ιδιαίτερα για την προαγωγή της σημασίας της ανάπτυξης υπαίθρου. Για τα μέτρα του πρασινίσματος, τα οικολογικά μέτρα τα λεγόμενα, θα ήθελα να ε, δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που έχουμε στο εσωτερικό των κρατών μελών για την προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα τα οποία λειτουργούν πολλές φορές ε, αποτελεσματικά και έτσι η ενίσχυση του οικολογικού ενδιαφέροντος ή η προαγωγή μέτρων οικολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ή να βάζουμε στο περιθώριο ή να παραγνωρίζουμε μέτρα και προόδους που έχουν ήδη επιτευχθεί στο εθνικό επίπεδο και γι' αυτό γεωργικά προγράμματα για το περιβάλλον που έχουν ήδη δώσει καλά αποτελέσματα, που έχουν επιστοποιημένα ε, επιτύχει θα πρέπει να συνυπολογιστούν ως μέτρα οικολογικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της νέας ε, μεταρρύθμισης για να φέρουν και τα αποτελέσματα τα επιδιωκόμενα και τα πλεονεκτήματα που άλλωστε ανέφεραν και οι συνάδελφοι νωρίτερα έχουμε πει στα θέματα του ελέγχου επί παραδείγματι και της επαλήθευσης για τα οποία θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια προς το συμφέρον των γεωγόρων μας και της υπαίθρου μας η ενίσχυση των μέτρων οικολογικού ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να ε, αποτελέσει μια εργασία ενίσχυσης της γραφειοκρατίας μόνο και διόγκωσης ε, ε, των γραφειοκρατικών μέτρων, αλλά είναι μια ουσιαστική ενίσχυση της διάστασης του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία θα ήθελα να δώσω εν προκειμένου στον, ορεινέ στις ορεινές ζώνες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και άρα με την ε, προσπάθεια για την ανάπτυξη υπαίθρου θα πρέπει να δώσουμε λύσεις αποτελεσματικές και ταυτόχρονα λύσεις οι οποίες θα είναι στο μέτρο της ε, τρέχουσας ε, οικονομικής κρίσης. Η ανάπτυξη πέθρου δεν μπορεί να αντέξει περικοπές, δεν θα πρέπει να εισεχθούν περικοπές οικονομικές. Θα πρέπει οτιδήποτε προσφέρεται να, έχει, να είναι σε ευθεία αναλογία με την πραγματική προσφορά του Γεωργού στην ύπεθρό μας, στη φύση μας και ελπίζω ότι έτσι όλοι μαζί με καλά μέτρα που θα εισαχθούν θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας μια επιτυχή μεταρρυθμίση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πάολος Κάρπατ, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Γερουσίας της Ιταλίας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πάολο. Ε, θα ήθελα να σου ανταποδώσω τις, ε, τους θερμούς χαιρετισμού σου και τα καλωσορίσματα ε, που έκανε στην αναρτήρια ομιλία σου. Η γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας έχει επανελειμμένως συζητήσει τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και μάλιστα έχουμε κάνει και ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα. Δεν υπήρξαν δηλαδή αποκλήσεις απόψεων ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες μέσα στην γερουσία μας. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο, Πρόεδρε, να υπάρξει μια πιο σαφής, ε, ένας πιο σαφής διαχωρισμός του πρώτου από το δεύτερο πυλώνα με το στόχο να ανταποκριθούμε στις απλου, απέτηση απλοποίησης ε, για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις αποσυνδεδεμένες άμεσες πληρωμές των ενεργούς αγρότες μειώνοντας όσο γίνεται το ποσοστό πολιτικής παρέμβασης. Επιπλέον το κάπινγκ θα μπορούσε τελικά να αποβεί ζημιογόνο ιδιαίτερα για κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, συνεργασίες ανάμεσα στους γεωργούς. Εν γέννη θεωρούμε πως η κατανομή της γεωργικής χρηματοδότησης ανάμεσα στα κάτι μέλη θα πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παράμετρο της επιφάνειας, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως ε, η παραγωγή, η προστιθέμενη αξία, το κόστος ζωής που διαφέρει από χώρα σε χώρα, η αξία της ε, γης αλλά και η ποιότητα και η ποσότητα της απασχόλησης που δίνει η γεωργία. Οι προτάσεις που γίνονται μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του, προϋπολογισμού για χώρες όπως η Ιταλία που θα ε, ε, ήταν θύμα μια τεράστια περικοπής που για μας είναι απαράδεκτο όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές. Πάντοτε για τις άμεσες πληρωμές θεωρούμε ότι το μίνιμουμ κατόφλι εξαίρεση που ισχύει για όλε τι χώρε θα πρέπει να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη απλοποίηση και οικονομία στην διαχείριση. Σε σχέση με το greening, η δέσμευση των ε, δικαιούχων γεωργών μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ισορροπία ε, ανάμεσα στι διάφορε παραγωγέ και χρειάζεται να προβλεφθεί μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβαση στα διάφορα κράτη-μέλη, πράγμα που θα ιδιολογείται από την απέτηση σεβασμού των διαφορετικών συστημάτων παραγωγή των διαφορών χωρών, αλλά και σε συμφωνία με τις αρχές της ενιαίας αγοράς και λόγω της ανάγκης να είναι λιγότερο ε, βαριά η γραφειοκρατία και ευκολότερη εφαρμογή. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο Βέλγιο, αλλά στην Ιταλία, όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, υπάρχει πραγματική ε, απέχθεια απέναντι στη γραφειοκρατία από πλευρά των Γεωργών. Ε, και σε σχέση με τις προτάσεις αυτές για μεταρρύθμιση θα πρέπει να κυριαρχεί το θέμα της γεωργικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας οι άμεσες πληρωμές χρησιμεύουν να ευνοήσουν τη γεωργική παραγωγή και ένα μεγαλύτερο ποσοστό αυτοανεφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δεν είναι αρκετά διευκρινισμένη η έννοια του ενεργού ε, αγρότη. Τώρα, σε σχέση με τα κυκλικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή λόγω της μεγάλης θετικότητας των βασικών ε, τιμών με τους αντίστοιχους κινδύνους για τα εισοδήματα, είναι απαραίτητο η μελλοντική γεωργική πολιτική να χαίρει συγκεκριμένων μέτρων για στήριξη των αγορών. Αλλά γι' αυτό βασιζόμαστε στις δικές σας ικανότητες και στη βούλησή σας. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα και εδώ κλείνω Προέδρε και εδώ θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ε, να δεχτούμε ως βασική παράμετρο την επιφάνεια Σα και μόνο. Ε, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε τους επιτρόπους που δουλεύουν πολύ καλά και επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω ε, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Λαβία για τη σπουδαία δουλειά που κάνει. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Σκάρπα και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Bundestag, Μίσερ Κόλμαν. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μα απευθύνατε. Με πολύ μεγάλη χαρά ήρθαμε. Συμμεριζόμαστε ανεπιφύλακτα τι προτάσει για την αναθεώρηση τη πολιτική και ιδιαίτερα του στόχου του. Τους στόχους της. Η Γερμανία είναι διατεθειμένη ταυτόχρονα να συζητήσει την ε, ανταγωνιστικότητα στην ε, Γεωργία, με τη νέα γεωργική πολιτική, την οποία πριν από τα άλλα κράτη-μέλη έχει θέσει σε εφαρμογή και μια πιο ανταγωνιστική παγκοσμίω ευρωπαϊκή γεωργία και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει ε, τις μεταρρυθμίσεις στον ίδιο δρόμο. Δεν θέλουμε οπισθοδρομήσεις, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Αυτό το απορρίπτουμε. Συμφωνούμε ιδιαίτερως ότι τα μέσα, τα κονδύλια στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να κατανέμονται καλύτερα και υπό την οπτική γωνία της ενίσχυσης των πιο, εκείνων που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ε, κοιτάξουμε και την ε, διάσταση του δεύτερου πυλώνα. Το κάπινγκ το απορρίπτουμε, δεν είναι, καμία, δεν λύση το να οριστούν όρια ανάλογα με το μέγεθο τη επιχείρησης. Η τωρινή λοιπόν γεωργική πολιτική είναι μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η κατάσταση στη χώρα μας. Η μετατόπιση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλών είναι μια λύση την οποία η πλειονότητα των μελών της αντιπροσωπείας μας, της επιτροπής μας απορρίπτει. Εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον μεταφορά κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο, εφόσον επιτρέπει πιο ε, καλή ασφάλεια στην υλοποίηση των μέτρων. Ειδικέ ρυθμίσεις όπως αυτές για τους νέους ε, γεωργούς ή για τους ενεργούς γεωργούς δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εισαχθούν και πάντως όχι πρακτικό να υλοποιηθούν. Εμείς θα είμαστε πίσω από κάθε μέτρο το οποίο θα οδηγήσει σε σωστή υλοποίηση του συστήματος. Δεχόμαστε τα μέτρα για την πράσινη κάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Dziękuję panu posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę pana posła σας τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καλινόφσκι. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι να αποκτήσει την νομιμοποίηση μεταξύ των ε, πολιτών. Έχουμε το πρασίνισμα, τα οικονομικά μέσα τα οποία πηγαίνουν στην ε, ΚΑΠ δεν θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτούς που δεν είναι αγρότες. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα εκείνο που έχει να κάνει με τις μικρές καλλιέργειες. Μιλάμε για τρία εκτάρια στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο μιλάει για πέντε δούμε τις μισές εκμεταλλεύσεις στην Πολωνία, αυτές είναι επιλέξιμες. Εντάξει, πρόκειται για μια απλοποίηση, για μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι κάτι θετικό, αλλά μόνο εδώ έχουμε να κάνουμε με απλοποίηση. Γιατί από την άλλη μεριά στη χώρα μου έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου οι μισές από τις μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις τελικά δεν ε, τις δουλεύουν οι ίδιοι οι αγρότες. Άλλοι τις ε, δουλεύουν. Οπότε τελικά αυτοί που δεν δουλεύουν στη γη θα παίρνουν ε, μια στήριξη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παίρνουν οι πραγματικά ενεργοί αγρότες. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν θα υπάρξει καμία ουσιώδης βελτίωση της κατάστασης. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη πρόταση στο θέμα των ε, άμεσων πληρωμών. Μα τελικά χρειαζόμαστε πάνω από 20 χρόνια για να ευθυγραμμιστούμε. Και μιλάμε για ισότιμους όρους. Νομίζω ότι στην πρόταση για το πρασίνισμα ίσως θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε και αυτό το κονδύλι για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για ορισμένες χώρες που περνάμε σε ενισχύσεις. Αν όλες οι χώρες δηλαδή έχουν την ίδια στήριξη για το πρασίνισμα, αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πιο δίκαιο από την σημερινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε και να ζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο Ευρωβουλευτής Ντόλ και μετά ο κύριος Κασικόφσκι. Παρακαλώ κύριε Ντόλ, έχετε το λόγο. Α, ο κύριος Ντόλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Σίγουρα ο εισηγητής κάνει πολλές προσπάθειες να δει στην πράξη τα διάφορα θέματα που αποσχολούν τις χώρες μέλη. Και σίγουρα πολλές ανησυχίες τις καλύπτει ο εισηγητής. Και εσείς κύριε Κάπουλο Σάντος με τις εκθέσεις σας έχετε προχωρήσει πολύ και έχετε βοηθήσει και την Ιρλανδία και στηρίξει στις θέσεις της. Στόχος βέβαια είναι η, η παραγωγή. Πώς θα γίνει βέλτιστη και πώς θα βρούμε το δρόμο μας ανάμεσα στους διάφορους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα πρέπει να φτάνουν στο στόχο τους. Σίγουρα εμείς εγκρίνουμε με πολλά από αυτά που προτείνονται από τους συγητές από των τεσσάρων ομάδων, από αυτά που άκουσα τουλάχιστον. Αλλά μια ερώτηση όμως έχω. Τώρα τι θα γίνει, θα εγκριθούν όλα αυτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ξέρω ότι 9 Ιουλίου λίγη προθεσμία. Μετά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν πρόκειται να εγκριθεί έτσι κι αλλιώς σύντομα μετά. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πού βρίσκεται. Πότε θα ολοκληρώσει και θα εγκρίνει τις εκθέσεις αυτές στα πλαίσια της συνολικής συμφωνίας, της φαιδικής συμφωνίας. Και πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα από τη δικιά σας την πλευρά για τη συνέχεια. Θα ήθελα να ξέρω και τις απόψεις των άλλων επιτροπών των ε, άλλων εθνικών κοινοβουλίων δηλαδή. Τι θα γίνει τελικά με την πρόταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουσικόφσκι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι γερουσιαστής. Εδώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε εδώ, που μας δώσατε την ευκαιρία να βοηθήσουμε και εμείς την εκπόνηση του πακέτου αυτού, όπως και οι συγητές. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε διάφορες λύσεις που για μας στη Γερουσία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά, πολλές αφιβολίες για το κατά πόσο πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Έχω δύο λεφτά στη διάθεσή μου, οπότε δεν θα μπω πολύ στις λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω τα Η γερουσία μας έχει ήδη παρουσιάσει τη θέση μας για το πακέτο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έχετε δηλαδή. Αλλά πιο συγκεκριμένα για τη θέση της γερουσίας και τη ε, διέτης, το θέμα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. η απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, η ανταγωνιστικότητα και η μη διάκριση όσον αφορά την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων στις διάφορες χώρες είναι για μας ζωτική σημασία. Ο κύριος Σάντος επέστησε την προσοχή μας το γεγονός ότι πουθενά δεν υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης σε βάρος κάποιας χώρας. Λοιπόν, εδώ θέλω να ξέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι τώρα δεν μας έχει απαντήσει. Είναι δυνατόν να υπάρξει διακριτική αντιμετώπιση των ε, χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να πρέπει να περιμένουμε 20 χρόνια για την ευθυγράμμιση. Αυτό δεν συνάδει με την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν τις χώρες, από όπου και αν είναι, Βαλκάνια ή αλλού ή την Πολωνία μπορείτε να μας μεταχειριστείτε διαφορετικά. Γιατί αν ναι, εντάξει. Αλλά αλλιώς ο πρόεδρος είπε ότι δεν θα ψηφίσουμε αν προηγουμένως δεν γνωρίσουμε τον προπολογισμό. Και είναι σωστό πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε λιγότερους σπόρους και περισσότερες απαιτήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Γερουσιαστά, τώρα ο κύριος Δησάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών που ε, έχω αναλάβει εκ μέρους της ομάδας μου την ευθύνη να ζητήσω μια παράταση για την κατάθεση των τροπολογιών. Δεν έχουμε το χρόνο δηλαδή να καταθέσουμε σε αυτά τα θέματα θα θέλαμε τις τροπολογίες μας να τις διατυπώσουμε και γι' αυτό παρακαλώ για την κατανόηση σας και μια μικρή παράταση. Θα πρέπει να λάβουμε μια ε, προσαρμογή στην κοινωνική πολιτική γιατί δεν μπορεί για τα ίδια προϊόντα ή ένα εκτάριο να παίρνουν ε, ε, διαφορετικά ποσά ο Λετωνός ή ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί ένας να παίρνει 78 και άλλος 550 ευρώ. Έτσι λοιπόν μεταξύ των 78 και των 550 ευρώ υπάρχει και η Ιταλία από ό,τι φαίνεται η οποία έχει εσωτερικές διαφορές από 50 ευρώ στην ενίσχυση για τον αγρότη στο νότιο Τυρόλο μέχρι 700 της Λομβαρδίας. Άρα λοιπόν καλό θα είναι πρώτα να κλείσουμε τη ψαλίδα στο ιστορικό των κρατών μελών και αναλόγως μετά να προχωρήσουμε για το greening, το πρασίνισμα. Πρέπει να σας πω ότι είμαι μάλλον ενοχλημένος από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι εισάγει πολύ περισσότερη γραφειοκρατία η πρόταση αυτή και δεν εξυπηρετεί τους στόχους της. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό της. 27 κράτη-μέρη δεν μπορούν να εισαγάγουν τα ίδια μέτρα για το greening. Άλλο η Φινλανδία, μα την δει κανείς από το αεροπλάνο, θα, έλεγα, θα έλεγε πού θα το βρει το 30% πρασίνημα πρασίνισμα. Αν πετάξει κανεί πάνω από τη Σικελία, θα πει ναι, το θέλει το 30% πρασίνισμα, αλλά που θα βρει το νερό. Ή πώ θα κάνει να πρασινίσουν ε, τα ηφαιστειογενή πετρώματα. Είναι πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ και ξέρω ότι πολλοί συναδελφοί στο Κοινοβούλιο ε, συμφωνούν μαζί μου. Χρειαζόμαστε ένα κατάλογο μέτρων ε, για το πρασίνισμα και βεβαίω αναλόγω θα καταθέσουμε και τι τροπολογίε μα ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο αυτό το οποίο σχέση με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν σημαντικά βελτιώσει οι συνάδελφοι εισηγητέ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο εκπρόσωπο τη Ισπανική Βουλή, ο κύριο Αλόνσο, έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Αλόνσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μέσα σε δύο λεπτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στις ανησυχίες μας σε σχέση με την πρόταση τροποποίησης για την κοινή γεωργική πολιτική. Πρώτο, όσον αφορά το θέμα του προπολογισμού. Η πρόταση του Ιουνίου του 2011 είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να δεχτούμε. Ο Πρόεδρος είπε ότι δεν θα υπάρξει τελική απόφαση αν προηγουμένω δεν έχουν αποφασιστική οι δημοσιονομικές προπτικές. Πολύ μας άρεσε αυτό. Και επειδή αν υπήρχε τροποποίηση του προπολογισμού, αν είναι προ τα πάνω τόσο καλύτερο, αν είναι προ τα κάτω όμως, αυτό θα σήμαινε μια αλλαγή στα έγγραφα αυτά και στις προτάσεις αυτές που εξετάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Τώρα το κείμενα του κυρίου καπουλεσάντου πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση πιστεύουμε. Θέλει ελαστικότητα όσον αφορά τα κριτήρια για τους ενεργούς αγρότες, τους μικρούς αγρότες, το πρασίνισμα τη παραγωγής. Τον ευχαριστούμε για τη δουλειά του. Όμως το πνεύμα της μεταρρύθμισης δεν αλλάζει. Λέει ότι τελικά ομοιογενώς πληρώνουμε για οικονομικές, κοινωνικές και αγροτικές καταστάσεις εντελώς διαφορετικές. Πράγμα που σημαίνει ότι αλλού θα πληρώνουμε χωρίς να πρέπει, αλλού θα χάνεται ανταγωνιστικότητα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω κύριε Κάπουλα Σάντος να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τα εκατομμύρια εκταρίων που θα εμφανιστούν ως ε, νέες εκμεταλλεύσεις στην κοινή γεωργική πολιτική. Αν είναι νέε, είναι γιατί πριν δεν ήταν γεωργικές οι εκμεταλλεύσεις αυτές. Ε, τι θα κάνουμε με αυτές. Και δεύτερον, τι θα κάνουμε με του τομεί εκείνου τη γεωργίας, ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, που παραδοσιακά είχαν οικονομική στήριξη, το γελαδινό γάλα και άλλα, που δεν συνδέονταν με μια γεωργική επιφάνεια μέχρι τώρα και κινδυνεύουν συνεπώς να χάσουν τις ενισχύσεις και άρα και την ανταγωνιστικότητά τους. Στον κύριο Νταντέν θέλω να πω ότι όσον αφορά την ενιαία οργάνωση αγοράς, αυτό είναι ένα στοιχείο ανησυχίας για τους αγρότες μας, γεωργούς και εκτινοτρόφους. Πρέπει, και εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος να το κάνουμε, να ζητήσουμε να έχει και πάλι η Ευρώπη ελαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία να μας επιτρέπουν σε πραγματικό χρόνο να αντιμετωπίζουμε την μείωση των τιμών, για όποιο λόγο και αν προκαλείται αυτή, και να υπάρχει ένα σύστημα τιμών αναφοράς που να βασίζεται στο κόστος της παραγωγής που να επιτρέπει την ενεργοποίηση τέτοιου είδους μέτρων. Εμείς στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι θετική η πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού στον αγροτικό τομέα. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο προκειμένου να ανακτήσουμε τις δυνατότητές μας για διαπραγμάτευση των ε, τιμών από πλευρά των γεωργών απέναντι στις ε, μεγάλες οργανώσεις διανομής των προϊόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπρόντφελτς. Labdien, priekšēdētāji kungs, cienītie kolēģi. Liels paldies σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση που έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε. Το Κοινοβούλιο της Λετωνίας παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση κοινωνικής πολιτικής. Εμείς θεωρούμε ότι, όπως υπόθηκε άλλωστε, οι άμεσες πληρωμές είναι η μεγαλύτερη αδικία, οι μεγαλύτερες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών εντοπίζονται στις άμεσες πληρωμές. Και ως εκ τούτου είναι και άθεμητος ο ανταγωνισμός. Οι τρεις βαλτικές χώρες από τη στιγμή που εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έλαβαν τις χαμηλότερες, τα χαμηλότερα επίπεδα αμέσων πληρωμών γιατί αυτές στηρίχθηκαν στα δεδομένα της περίοδου 94 με 99 και ήταν ήδη πάρα πολύ χαμηλές. Στην περίοδο εκείνη 94-99 είχαν το χαμηλότερο επίπεδο επίπεδο, στη γεωργική του παραγωγή, αλλά γενικότερα στην οικονομική του δραστηριότητα οι χώρε αυτέ, οι τρει βαλτικέ χώρε, διότι είχαν μόλι βγει ε, από μία περίοδο καθεστώτος ε, μη ελεύθερης αγοράς και έκαναν την μεταλλαγή στην ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπολογιστούν με νέο τρόπο αυτές οι άμεσες πληρωμές για τις ε, χώρες μας και με διαφορετική χρονική περίοδο αναφοράς. Θα πρέπει να υπάρξει ισότιμη κατανομή των ποσών των αμέσων ε, πληρωμών και να πάψουν οι μεταβατικές περίοδοι. Μπορεί να προβλέπετε το 65% ε, επί του μέσου όρου των άμεσων πληρωμών για κάθε γεωργό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτελεί ήδη ένα βήμα προ την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι επαρκέ και δεν το δέχεται ω εκ τούτου η Λετωνία, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 80% του μέσου όρου, επί του μέσου όρου των άμεσων πληρωμών να εισπράττει ο κάθε γεώργο για να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα αυτό θα φέρει για τι χώρε τη Βαλτική το ποσοστό του 80% επί του μέσου ορού άμεσων πληρωμών, θα χρειαστούμε ακόμη 2,1 δις ευρώ, ποσό μηδαμινό, 0,71% μόνο επί του ε, κοινοτικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισότιμες άμεσες πληρωμές, δίκαιες, ισοδίκαιες και Διαφορετικά θεωρούμε ότι θα ήταν ίσως ακόμη πιο ισότιμη η κατάσταση αν δεν υπήρχαν καν άμεσες πληρωμές. Αλλά πάντως όχι τώρα με το σύστημα που έχουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάιον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν και εισηγητής, όπως και ο κύριος Ντέ, Έχετε το λόγο κύριο Λάιον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους φίλους ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθαν εδώ για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Και θα ήθελα ξεκινώντας να υπενθυμίσω ότι η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν είναι ένα τετριμένο γεγονός πλέον, διότι μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας υπάγεται πλήρως τη διαδικασία της συναπόφασης κοινή γεωργική πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να αναλάβει πλήρως το ρόλο που του ανήκει στη διαδικασία αυτό. Γι αυτό, αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες από τις ανησυχίε που ενδεχομένω εκφράζονται ως προς την ε, μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και, την, ε, και τις θέσεις που μπορεί να έχουν εκφραστεί επίπεδο Συμβουλίου ή πώς μπορεί να τις προβάλλει η Προεδρία της Δανίας μες στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς θα απαντήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφέ τι περιμένουμε και τι αναμένουμε από την υπόθεση αυτή. Η συναπόφαση δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αποφάσεις που θα λάβουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μέσα στη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφέ. Ε, η κοινή γεωργική πολιτική λοιπόν θα πρέπει στη μεταρρύθμισή της να χαρακτηριστεί και από λιγότερη άντληση ενεργειακών πόρων αλλά και λιγότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη η γεωργία που θα προκύψει μετά την ε, μεταρρύθμιση αυτή, μετά την αναθεώρηση αυτή. Και οι ανησυχίε που εκφράζουν πολλοί συνάδελφοι άλλωστε στην Επιτροπή Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι ορισμένε από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον προ τα πίσω μα πηγαίνουν παρά προ τα μπρο και ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο τελικός στόχος της ε, διαδικασίας αναθεώρησης. Ειδικότερα δε στο θέμα του, των μέτρων οικολογικού ενδιαφέροντος, του greening δηλαδή, υπάρχει σαφέ ενδιαφέρον από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάσκεψη τη οικολογικότερη παραγωγή. Ωστόσο, οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίε έχουν ένα χαρακτήρα ομοιόμορφο και τείνουν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, τα τρία αυτά μέτρα τα οποία επιτεθούνται εφαρμόζονται απανταχού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω χωρί να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερε ανάγκε και ιδιαιτερότητε ε, στα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε, θα πρέπει να ε, αναθεωρηθούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θεσπίσει με τι ε, ψηφοφορίε του νέε ρυθμίσεις, με τις τροπολογίες, έτσι ώστε να επιτρέψει τα καράτη μελη μια διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με την ε, περιοχή. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στη βιοπικιλότητα, που είναι επίση βέβαια πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να εστιάζονται και στην αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και την αποτελεσματικότητα στην ε, και, και τον περιορισμό μάλλον των εκπομπών ε, άνθρακα που είναι σημαντική και κοινική στόχη. Ελπίζω λοιπόν ότι από κοινού και μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε τους στόχους αυτούς γιατί βλέπω ότι όλοι συμφωνούμε. Επίσης ε, η κύρωση για την αποτυχία στην προσπάθεια για μια διάσταση οικολογικότερης παραγωγής θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια η άμεση πληρωμή. Αυτό θα πρέπει να είναι το τίμα που θα πληρώσει κανείς αν αποφασίσει να μην υλοποιήσει τα μέτρα για την οικολογικότερη παραγωγή. Επίσης όσον αφορά νέους, ε, ε, νέους δικαιούχους, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη ακόμη χρησιμοποιούνται ιστορικά, ιστορικές αναφορές για τις ε, πληρωμές, η ταχύτητα και τα βήματα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζονται τροποποίηση και θα θέλαμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Η Αυστρία παρακαλώ. Τώρα ο εκπρόσωπος του Αυστριακού Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, θα θέλαμε και εμείς μια γενική ε, ο κύριος Έσλ. Θα θέλαμε μια καλή γεωργία, μια γεωργία η οποία, μια μεταρρύθμιση γεωργικής πολιτικής η οποία θα φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι αποδεκτή η δεν είναι αποδεκτή διαχωρισμοί μεταξύ ε, πλεονεκτούντων ε, και μη πλεονεκτουσών και μη εκτάσεων. Οι κτηνοτροφικέ επιχειρήσει, παραδείγματι, για τις ορεινέ περιοχές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν ε, επίση ε, ε, επιχειρήσει οι οποίες χρειάζεται, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που ισχύουν, να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο και ενδεχομένως ε, να προστατευτούν με περισσότερη, υψηλότερες άμεσες πληρωμές, γιατί διαφορετικά θα μπορούν να συντηρηθούν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ως προς τις ε, αλπικές ζώνες και τις γεωργικές μεταλλεύσεις που βρίσκονται εκεί. με πολλές δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε Εάν υπάρχουν 100 εκτάρια και άνω σε μια γεωργική εκμετάλλευση και 30% εξ αυτών είναι ε, λιμόνες ε, τουλάχιστον το καλοκαίρι, να θεωρούνται άμεσα και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες ως ε, μέτρα οικολογικότερης παραγωγής, ως πρασίνισμα δηλαδή. Για το πρασίνισμα επίσης, η διατήρηση των, ε, των πράσινων εκτάσεων δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή για την εκμετάλλευση εκεί όπου βλέπει ότι έχει μεγαλύτερο περιθώριο για πράσινη έκταση να το αξιοποιεί, να μην είναι υποχρεωμένη δηλαδή πάντοτε να έχει την ίδια αναλογία. Επίσης το σύστημα με τους ελέγχους για μένα είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα Η κυρία Όσκαρσον. Σας ευχαριστώ, θα τα πω σου ειδικά. Σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε. Ε, έχω ακούσει με πολύ προσοχή όλους τους συναδέλφους. Ήδη νομίζω γνωρίζετε τη θέση της Σουηδίας ε, για το θέμα αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ε, ισχυρός ε, προϋπολογισμός, ο οποίος όμως να χρησιμοποιηθεί και αποτελεσματικά, ώστε να αποδώσει, είναι σημαντικό ο γεωργικός τομέας ε, να είναι αποδοτικός, να βοηθηθεί με αποτελεσματικά μέτρα, όπως το greening, το πρασίνισμα. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο περιεχόμενο και ο συγκεκριμένος κοινό ορισμός για τις διάφορες χώρες, ε, κοινοί κανόνες για όλους όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να ε, γίνεται επίσης όρις ο ανταγωνισμός. Είναι σημαντικό ο δεύτερος πυλώνας να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό είναι θετικό και για τους νέους αγρότες που θα μπορούσαν να βοηθηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί θα πρέπει να διευκολυθούν ώστε να εγκαταλείψουν την παραγωγή, να αφήσουν το επάγγελμα με κάποιο τρόπο Έχουμε μια γενική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στη γεωργία το ίδιο, με περισσότερο πρασίνισμα, ε, πιο αποτελεσματικό χρήσο των πόρων ε, και είναι σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια και όσον αφορά τη στήριξη των ε, μειονεκτουσών περιοχών. Δεν συμφωνώ με τον αυστριακό συνάδελφο θα πρέπει να βρεθεί, ε, θα βρεθούν λύσεις και για τις ορεινές ή μειονεκτούσες περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκαρθία. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ που οργανώνεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με τους εθνικούς βουλευτές. Επίτα, θέλω να πω μερικά πράγματα για τους στόχους πέρα από την εφαρμογή. Δηλαδή, το θέμα είναι μερικές φορές το πώς, αυτό που κάνουν πολλές φορές είναι ότι κοιτάνε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες της κοινή γεωργικής πολιτικής, ενώ μερικές φορές πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι στόχοι τη γεωργικής πολιτική είναι σωστοί. Ο στόχο είναι να υπάρχουν αρκετέ ποσότητε τροφίμων σε καλέ τιμέ και σε καλή ποιότητα. Αυτό είναι ο στόχο. και αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε. Από εκεί και πέρα υποστηρίζουμε ότι ο πρωτογενή τομέα είναι στρατηγική σημασία, όπω και η ενέργεια, όπω και η άμυνα, όπω και η ασφάλεια. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Ο προπολογισμό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμω θα πρέπει να δούμε και άλλα. Η πρόταση εδώ είναι καλή που δίνει την ελευθερία στις χώρες μέλη να αποφασίσουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Υπάρχουν θέματα όπως είναι η κτηνοτροφία ε, των κοινών που δεν έχει λυθεί. Είναι θέμα επίσης των δεδεμένων ε, ενισχύσεων. Αλλά αν όλα τα βάλουμε σε αυτές τις ενισχύσεις θα ήταν τραγωδία αυτό για πολλούς παραγωγούς. Συμφωνώ με τους συναδέλφους από το ΕΛΚ ότι το πρασίνισμα δεν μπορεί με τον ίδιο τρόπο να εφαρμοστεί παντού, ούτε τα μέτρα μπορεί να είναι ίδια σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γεωπονικές διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για την ε, ενοποίηση των, ε, ε, της βοήθειας από τον πρώτο πυλώνα. Πρόκειται για την απώλεια εσόδων για τους αγρότες και για ποιου λόγους. Για συγκεκριμένου λόγους. Υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχει η προστασία των κτλ. Υπάρχει και ένα δεύτερο, το οποίο έχει άμεση σχέση εδώ και είναι οι συμφωνίε που έχουμε υπογράψει και με τι συμφωνίε αυτέ αυτό που κάνουμε είναι ότι αφαιρούμε ανταγωνιστικότητα από του αγρότε μα. Και αυτό το δεύτερο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Όσο δεν έχουμε ε, δημοσιονομική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε όλο και περισσότερε χώρε μέσα στο ευρώ, δεν είναι δυνατόν ομοιογενώ να εφαρμόζουμε την κοινή γεωργική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, το πιο σημαντικό για κάποιου τομεί και δεν έχει συζητηθεί αυτό ακόμα σήμερα, είναι οι ενισχύσει των αγορών, οι οποίε αναφέρονται στην έκθεση Νταντάν. Και γι' αυτό και η πρόταση Νταντάν είναι πάρα πολύ σημαντική και θα προσπαθήσουμε να την βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο με τροπολογίε, αλλά είχε πολύ θάρρο ο κύριο Νταντάν με τι προτάσει που παρουσίασε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκπρόσωπος της Ρωμανίας, ο κύριος Αντουλέσκου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις προσπάθειές τους σε σχέση με αυτό το πακέτο. Όσον αφορά την θέση της Ρουμανίας, και την προστασία των φυσικών πόρων και την ε, μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει να σας πω τα εξή. Η Ρουμανία υποστηρίζει το γενικό επίπεδο των επιχορηγήσεων για την ε, κοινή γεωργική πολιτική που προτείνει η Κομισιόν. Είναι το μήνυμο που θα μπορούσε να αποδεχτεί η Ρουμανία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι εθνικοί προβληματισμοί. Καταρχήν, η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Η Ρουμανία θα ήταν υπέρ ενό ενιαίου ποσοστού, γιατί η υπολογισμοί σύγκληση που προτείνει η Κομισιόν διατηρεί την διαφορά ανάμεσα στο μέγιστο και στο μήνυμο επίπεδο που χορηγείται στους, στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η, η οροφή της στήριξη που δίνεται στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Είμαστε κατά. Τρίτον, η το πρασίνισμα των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο για τους γεωργούς. Άρα λοιπόν το ποσοστό της 30, του 30% των άμεσων πληρωμών είναι εξαιρετικά υψηλό. Εμείς θέλουμε δύο διαφορετικές οροφές. Ε, ένα, ε, μία για το εισοδήματα των γεωργών, για τις άμεσες ε, πληρωμές δηλαδή, και ένα άλλο ανώτατο όριο για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές που θα πρέπει να είναι επίσης τα ίδια ποσοστά για ολόκληρο ολόκληρη την Ευρώπη. 20% δεν είναι το όριο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου δε, η Ρουμανία θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους και το βάρος αυτού του δίκτυ θα πρέπει να υπολογιστεί στον υπολογισμό της κατανομής των πόρων. Όσον αφορά τώρα την συγχρηματοδότηση, εμείς δεν υποστηρίζουμε το ποσοστό 4%. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ισχύσει το 7% και μάλιστα ποσά τα οποία θα μπορούν να είναι μεταβιβάσιμα σε δύο φορές. Όσον αφορά τις ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εφαρμοστούν με διαφοροποιημένο τρόπο. 3% για τις εκμεταλλεύσεις μέχρι 20 εκτάρια και 5% για τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, δηλαδή άνω των 20 εκταρίων. Στη συνέχεια θα πρέπει επίσης να γίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη, γιατί τα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρδευση, η άρδευση είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της παραγωγής αυτών των νέων κρατών μελών, όπως και η Ρουμανία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, κύριος Μπατίστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Συμφωνούμε για την κοινή γεωργική πολιτική και το γεγονός ότι αποτελεί την βασική εγγύηση για την ε, ανεφοδιασμό σε τραύμα. Είναι ωστόσο σημαντικό να προστατευτεί η φύση αλλά και η χωροταξία. Και εδώ πιστεύουμε ότι ένα τμήμα της ε, γεωργίας της είναι και η καινοτομία αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν αρκεί όμως να μιλάμε για όλα αυτά. Θα πρέπει να ληφθούν παρετέρω μέτρα τα οποία να είναι λειτουργικά. Ω εκ τούτου θεωρούμε ότι η έκθεση την οποία συνέταξε ο βουλευτής Καπούλα Σάντος και τον ε, θαραλέο τρόπο με τον οποίο ε, προσπαθεί να προτείνει μέτρα και να τα θέσει και σε εφαρμογή ε, τα μέτρα τα οποία προτείνει στους γεωργούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα κοινό, ένα κοινό στόχο που θα είναι η σύγκληση της τάξης του 80 με 90%. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν, θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια πραγματική συνένεση, ώστε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επικράτεια να τη χάνει του ίδιου επίπεδου στήριξης, αντίστοιχο με την ε, γεωργική παραγωγή και ε, ικανό ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη της υπέδρου. Έχουμε μια πρόταση ιδέα ε, που έχει να κάνει με το greening, το πρασίνισμα της κοινή πολιτικής είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο κατά τη γνώμη μας ε, δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε τα σχετικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή όσον αφορά τις πολιτιστικές διαφορές και τις συνθήκες που ισχύουν στις μεσογειακές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα το θέμα της άρδευσης. Στις μεσογειακές περιοχές δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ένα επίπεδο παραγωγής και ικανοποίησης όσον αφορά το καθεστώς greening, εάν δεν υπάρξει στήριξη για την ε, άρδευση. Επιπλέον πιστεύουμε ότι το greening θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο και όχι ως ποινή. Να εκφράσουμε λοιπόν ε, τη λύπη μας που η έκθεση της Κομισιόν δεν έχει ορίσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για τη σύγκληση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα στήριξης για τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μάρτιν Ροστίνγκ, ζητώ συγγνώμη και πάλι. Ναι, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας καλωσορίσω καιρό και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουν μόνο συντηρητική δικαίωμα λόγου στην αίθουσα αυτή, αλλά και εμείς. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στην διάσταση οικολογικότερη παραγωγή, γιατί είναι η πιο απαραίτητη και η πιο σημαντική μεταρρύθμιση. Και ο κύριο λόγο πλέον για άμεσε πληρωμέ στη νέα περίοδο. Υπάρχει μια προσπάθεια για ευέλικτη οικολογική παραγωγή ή και για πλήρη καταργησή της. Αυτή όμως θέτει σε μεγάλο κίνδυνο και τους παραγωγούς στο σύνολό τους. Και εμείς πιστεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να ε, υπάρχουν αυτές οι βάσεις για την διάθεση των ενισχύσεων στη γεωργική παραγωγή. Το λέμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο το λέω ξεκάθαρα, χρειάζεται νέα και πιο δίκαιη κατανομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν, αλλά και καλύτερη κατανομή μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε στη μεταρρύθμιση και επίσης σημειώνουμε ότι δύο τρίτα του Κοινοβουλίου έχουν υποστηρίξει το capping, το όριο μεγέθους δηλαδή επιχείρησης. Δεν υπάρχει λόγος ε, να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει του αντίο να επικεντρωθούμε στις μικρότερες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το δεύτερο πυλώνα προβλέπεται το 30% για την για τα οικολογικά προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας ενιαίος στόχος και ένα νέο μέτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα λόγο να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις τη υλοποίηση τους. Αλλά σε στόχος θα πρέπει να υπάρχει. Και ένα πράγμα που δεν χρειάζεται δεύτερος πυλώνα είναι η πρημοδότηση της ε, εγκατάλειψης τη παραγωγής για τον ε, παραγωγό. Δεν υπάρχει κανένας λόγο να χρηματοδοτούμε τους παραγωγούς και να σταματήσουν να παράγουν. Άρα τα ποσά αυτά θα πρέπει στον πρώτο πυλώνα να πάνε ή στο ειδικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερα υποστηρίζω τις προτάσεις του κ. Νταντά. Χρειάζονται ε, προτάσεις ε, για την οργάνωση αγοράς, όχι μόνο για τον ίνο ή για τη ζάχαρη, αλλά και για άλλα προϊόντα. Και καλό τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια να ξανασυζητήσουν το θέμα του γάλακτος. Η κρίση στη γαλακτοπαραγωγή μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά μέτρα και με ποσοστώσεις, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγορά γάλακτος. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον κανόνα. Τώρα θα έχουμε τρεις εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και έναν Ευρωβουλευτή κάθε φορά και θα ήθελα για ακόμη μια φορά να σας ζητήσω να σεβαστείτε το χρόνο που σας έδωσα δύο λεπτά έκαστος. Ο κύριος Νέγκρη από το Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη σημερινή πρόσκληση. Η κοινή γεωργική πολιτική δίνει έμφαση σε ένα εντονότερο πρασίνισμα. Για την ώρα πρόκειται για το 7% των αρρώσιμων γεών με υψηλή οικολογική αξία. Ο κύριος Κρίστενσεν πριν από λίγο πρότεινε η πληρωμές να μειώσουν το ποσοστό αυτό στο 3,5% εάν ληφθούν ε, και άλλα επιπλέον μέτρα. Όντως αυτό το ποσοστό 7% είναι σχετικά ψηλό. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει περισσότερο να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια, πάντοτε με στόχο ένα πιο έντονο πρασίνισμα. θα πρέπει ίσως να μείνει το 7% μόνο για τις ζώνες υψηλής ε, οικολογικής αξίας. Θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πίτερς θα πάρει το λόγο τώρα. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Μου είπανε δύο λεφτά για το πρασίρισμα. Η γεωργία χρειάζεται βέβαια πολύ χώρο, ε, πολύ γη. Η ποιότητα όμως τα τελευταία χρόνια πάει πίσω και υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ε, σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκεται το έδαφος. Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν πάει καλά η ποιότητα του εδάφους. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ποιότητα των ε, εδαφών για να πετύχουμε ένα μοντέλο τροφίμων που θα μας προσφέρει τρόφιμα ποιότητας που το χρειάζεται τόσο πολύ ο κόσμος. Χρειάζεται λοιπόν βιώσιμη γεωργία, που σημαίνει ότι χρειάζεται οικολογική παραγωγή. Πολύ βασικό και για να το πετύχουμε αυτό για μας, στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς η γεωργία πρέπει να καλύπτεται από τα αναγκαία μέσα. Βέβαια είναι ειδικό το πλαίσιο που έχουμε στη Φλάνδρα πρέπει να ξέρουμε. Γιατί υπάρχει κατακερματισμένη γη και οι τιμές των, ε, της γης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Η γεωργία γίνεται συχνά ε, στις περιαστικές περιοχές και εκεί υπάρχει κατακερματισμός ο προπολογισμό του να μπορεί να πηγαίνει από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 για μα είναι πολύ θετικό. Αλλά επανέρχομαι λίγο στο θέμα του πρασινίσματος. Υποστηρίζεται απόλυτα ε, να υπάρχει μια πιο οικολογική παραγωγή και οι άμεσες πληρωμές πάνε προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτός είναι ένας αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει αποτελεσματικός χωρίς να πληγεί όμως η απόδοση ή χωρίς να πληγεί το περιβάλλον και η φύση. Χρειάζονται ειδικά μέτρα για την κάθε περιφέρεια, για την κάθε περιοχή, για να επιτευχθεί ο στόχος του πρασινίσματος. Θέλουμε η Ευρώπη να διατυπώνει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την περιφέρεια και χωρίς όμως να αυξηθεί η γραφειοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ελαστικότητα ώστε κάθε η περιοχή να μπορεί να προσαρμόζει τα μέτρα ανάλογα με τις ιδιαιτεροιότητες της. Και αυτό να ισχύσει και στο πρασίνισμα και στην αϊφόρο γεωργία γενικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο ομιλίας και τώρα ο κύριος Πανικέβεν. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας απόγευμα. Όντως, είμαι από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και θέλω να υπογραμμίσω 7 σημεία όσον αφορά την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής. Όντως θέλουμε να ενισχύσουμε την κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε δίκαιες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Εμείς στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι η έρευνα είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και το 10% για την ε, γεωργική παραγωγή σημαίνει για μας κάπου 30 δισεκατομμύρια να πηγαίνουν στην έρευνα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι θα υπάρξει αποσύνθεση όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα για το πρασίνισμα. Ένα άλλο σημείο είναι ότι εμείς δεν θέλουμε η στήριξη η οποία δίνεται να συνδυάζεται με την παραγωγή. Γιατί αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Ένα άλλο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι για όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες της υπονάπτυξη χώρες και να κάνουμε και μια εξολόγηση αντικτύπου. Έκτο σημείο έχει να κάνει με την ανακατανομή των μέσων. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένες χώρες παίρνουν περισσότερα από άλλες, αλλά για την Ολλανδία αυτό σημαίνει 8% περισσότερο από ό,τι δίνουν άλλες πλούσιες χώρες. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Και τέλος, Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω ότι και εμείς είμαστε υπέρ της μείωσης της γραφειοκρατίας όσο γίνεται περισσότερο. Είναι γνωστό ότι στην απλοποίηση υπάρχει και η αξία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Πόλσεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ εργάζομαι κυρίως με τα γεωργικά προγράμματα και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε αυτό το θέμα στην παρέμβασή μου. Ο Κάπουλα Σάντος έχει γίνει διάσημος γιατί πραγματικά πρόσεξε και έλαβε υπόψη τις διάφορες απόψεις που εμείς του υποβάλαμε ως σκιώδεις εισηγητές στην έκθεση του για παράδειγμα τώρα στο κείμενο του Συμβουλίου και της Κομισιόν γίνεται λόγος για ευημερία των ζώων ως ε, μία από τις προτεραιότητες. Για μένα αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ε, υπάρχει και συμπεριλαμβάνεται και ο αγροτοτουρισμός. Αλλά εσείς που δουλεύετε σε εθνικό επίπεδο, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Όλη αυτή την περίοδο μιλήσαμε για θέματα περιβαλλοντικά, για το περιβάλλον και είναι προφανές ότι αυτό είναι βασικό για την επιβίωση του είδους μας. Αν όμως θέλουμε να διατηρήσουμε μια γεωργία ζωντανή, Στι στις χώρες μας, μια γεωργία ε, που θα είναι και η προϋπόθεση για μια ζωντανή και αναζωογονημένη κοινωνία θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε σε περιβαλλοντικό και επίπεδο να υπάρχει δυνατότητα να ζει κανείς καλά στην εξοχή, στην Ήπεθρο. Όχι μόνο η γεωργία αλλά και όλοι όσοι ζουν στην Ήπεθρο. Όταν λοιπόν συζητάμε για αυτά τα θέματα γεωργίας, ε, του γεωργικού, του χώρου, της Ήπεθρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ζωντανή Ήπεθρος είναι απαραίτητη απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και τη συνέχιση της γεωργίας μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη, όχι μόνο μέσω της γεωργίας και της δασοκομείας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κούπης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριος Πουπίνης. Και ευχαριστώ πολύ και τους εισηγητές και του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητούμε σήμερα και υποστηρίζουμε πολλέ από τι τοποθετήσει που ακούστηκαν για τη μεταρρύθμιση τη κοινή ε, γεωργική πολιτική, πολλέ από τι θέσει τη μεταρρύθμιση για το, για το θέμα των άμεσων πληρονομών όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι καθόλου ε, ίση η κατανομή των εσόδων μεταξύ γεωργών ε, στην Ευρώπη και των άμεσων ε, πληρωμών, ειδικά όσον αφορά τα τρία βαλτικά κράτη, Λιθουανία, Λετωνία και Εστονία. Υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και περιμένουμε μέτρα στήριξη για την εξουσία των άμεσων πληρωμών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που κατέθη σήμερα έχει να κάνει με τις ε, γεωργικές και εκτάσεις και την ε, απογραφή τους. Είχαμε επί 50 χρόνια εθνικοποιημένες ή κρατικοποιημένες εθνικές γέες, τώρα όμως επανέρχονται στα χέρια των νόμων κατόχων τους. 2,6 εκατομμύρια εκτάρια δηλαδή γεωργικών γεών επανέρχονται στα χέρια των νομών ε, δικαιούχων και θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα του πώς θα υπολογιστούν οι άμεσες ε, ενισχύσεις για αυτές τις ε, επιφάνειες, τις εκδάσεις. Επίση, το θέμα τη ανάπτυξη τη υπαίθρου είναι διαφορετικέ οι ανάγκε και δεν είναι δυνατόν ε, να περικοπούν ε, οι ε, ενισχύσει στην στιγμή που παλαιότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σχεδόν τέλειες υποδομές, έχουν να αξιοποιούν την νέα τεχνολογία, ενώ χώρες όπως οι δικές μας δεν έχουν τέτοιες ευκαιρίες, ούτε είχαν τις ευκαιρίες στο παρελθόν πρόοδο δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε χωρί την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει, πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τι άμεσε ενισχύσει. Εκεί πρέπει να ζητήσουμε καλύτερε λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκπρόσωπο ε, τη βουλευτή από τη Φιλανδία, ο κ. Σέτανεν. κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις της Κομισιόν και το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής είναι μια σωστή βάση για διαπραγματεύσει. Ωστόσο θα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν οι προτάσεις και να απλουστευτούν οι προτάσεις. Ε, ωστόσο, ε, συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε τις συνδεδεμένες πληρωμές για παραγωγή υπό τις δικές μας συνθήκες. Πρέπει να αλλάξουν οι απαιτήσει, οι όροι ωστόσο για να ληφθούν υπόψη διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να, την γεωργία. Ε, το πάνω από το 60% της επιφάνειας της Φιλανδίας θεωρείται ως ε, φυσική, περιοχή με φυσικά μειονεκτήματα. Αυτό θα πρέπει να ε, συνεχίσει να ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το κόστος μέσω των επενδύσεων των γεωργών. Το ο, καιρό. Επίσης έχουμε σοβαρή ανησυχία όσον αφορά την άρση των ποσοστώσεων, την κατάρριση των ποσοστώσεων. για την ζάχαρη θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το 2020 και ακόμα και πιο μετά γιατί διαφορετικά η μόνη μας βιομηχανία ε, στη Φιλανδία κινδυνεύει. Για τη Φιλανδία είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η σημερινή δυνατότητα συγχρηματοδότησης, όπου το κοινοτικό τμήμα μπορεί να φτάσει από το 25 μέχρι το 75% για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Φιλανδία χρησιμοποιεί πολύ εθνική συγχρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να διαφέρει... Ε, και να λειτουργήσει διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης έχουμε συζητήσει στη Φιλανδία ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πλήρη συμμετοχή στην ε, επιστροφή από την αγορά. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Εστονίας, ο κύριος Κόβα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, με χαρά ακούω σήμερα ότι πολλοί από εσά έχετε ήδη αντιληφθεί τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν λόγω των μεγάλων αποκλήσεων στι άμεσε πληρωμέ στα βαλτικά κράτη. Ελπίζω ότι με τη δική σα βοήθεια θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να στηρίξουμε τα ε, κράτη-μέλη ε, που της Βαλτικής ε, σε αυτή την προσπάθεια να βελτιώσουν το επίπεδο των γεωργών τους. Η πρόσθετη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα επιτρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη για δραστηριότητες που δεν προσθέτουν προσθέμενη αξία ή στο περιβάλλον ή στην κοινωνία. Ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι όταν ε, μιλάμε για μια προσθέμενη αξία για την κοινωνία θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις λύσεις που ήδη έχουμε εντοπίσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και πάνω απ' όλα ευχαριστώ για τη συντομία σας. Ο κύριος Γιάννη Βοησντροφσκή, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να σας πω τίποτα καινούριο εδώ μέσα, γιατί έτσι κι το πρόγραμμα στο οποίο θα αναφερθώ το έχουν αναλύσει και οι συνάδελφοι μεταξύ άλλων και ο κύριος Πουπίνης από την Λιθουανία. Όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε μία προφανή διάκριση. Είναι μια διάκριση η οποία απορρέει από μια ανισότητα όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές. Έχει γίνει έκκληση να χρησιμοποιηθεί ο ρεαλισμός. Αυτό ζητήσαμε εδώ στην αίθουσα. Οι συνάδελφοι από τις χώρες που έχουν τις πιο χαμηλές άμεσες πληρωμές πρέπει να εφαρμόσουν τον ρεαλισμό. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Η έκκληση αυτή θα ήταν ίσως πιο εύκολη αν ήταν μόνο οικονομικό το ζήτημα. Δεν είναι όμως μόνο οικονομικό. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Οι νέες χώρες μέλη, γιατί είναι κυρίως οι χώρες, ε, οι καινούργιες μέλη που πλήττονται, σε αυτές λοιπόν γίνεται μια διάκριση όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Εμείς θέλουμε να μην γίνεται διάκριση για καμία χώρα. Χώρες όπως η Πολωνία ή η Λιθουανία παίρνουν λιγότερα χρήματα. Και όχι γιατί δεν τηρούν τα κριτήρια, αλλά επειδή οι εκμεταλλεύσεις τους είναι ακριβώς από αυτές τις χώρες και όχι από άλλες. Μα αυτό είναι απαράδεκτο. Ακόμα δεν έχει απαντήσει κανείς. Εγώ αυτό το θέμα το έχω θίξει πολλές φορές μέχρι σήμερα και δεν έχω πάρει κανένα νομικό επιχείρημα το οποίο να δικαιολογεί μια τέτοια κατάσταση. Γίνεται λοιπόν μια διάκριση σε βάρος των νέων χωρών. Δεν γίνεται όμως γιατί αντιβαίνει στις ίδιες τις συνθήκε. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να παίρνουν περισσότερα επειδή πάντοτε στο παρελθόν παίρναν περισσότερα και κάποιοι να παίρνουν λιγότερα επειδή πάντα παίρνανε λιγότερα. Αυτό το ιστορικό κριτήριο είναι άδικο και αντιβαίνει στις συνθήκες και ούτε μπορεί να σταθεί νομικά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βρούμε μια νέα λύση που να είναι ρεαλιστική πολιτικά αλλά και να τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί να παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο και να εφαρμόζουμε αρχές οι οποίες αντιβαίνουν στην αρχή της μη διάκρισης. Πρόεδρος, ο κύριος Βοητσοχόφσκι είναι δικηγόρος. Οφείλω να σας το πω αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Χόφκιν από τη Γερμανική Βουλή. Κυρία, και σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χόφκιν, για την ε, πολύ καλή συνεργασία με όλες και όλους τους συναδέλφους. Πιστεύω θα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για έναν προϋπολογισμό ισχυρό για ένα καλά εξοπλισμένο ε, γεωργικό εξοπλισμό. Αυτό τουλάχιστον το επιδιώκουν και τα δύο σώματα της Γερμανικής Βουλής ε, και το Bundestag και το Bundesrat και πιστεύουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από την σημασία του που θα αποδοθεί στον προπολογισμό Τη γεωργίας και στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Επίσης, ο επίτροπο Γεωργίας κ. Τσόλο μας έχει κάνει κάποιες προτάσεις γιατί ο πρώτο πυλώνα όπου το Bundesrat έκανε συγκεκριμένες προτάσεις και θα ήθελα επί την ευκαιρία να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον κύριο Καπούλο Σάντος που τις έλαβε υπόψη του. Ιδιαίτερα για τα όσπρια. Και επίσης η έκθεση της κυρίου Νταντέ μου φαίνεται πολύ σημαντική, διότι θα πρέπει στις εποχές που διανύουμε να μιλήσουμε λησμονούμε πόσο σημαντικό είναι να προχωρούμε και στην αναθεώρηση ε, ορισμένων μέτρων απορρίθμισης. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη, για τη χρηματοπιστωτική αγορά, αλλά και για τις ε, οργανώσεις αγοράς. Άρα λοιπόν, και στη Ζάχαρη, αλλά και σε άλλες οργανώσεις αγοράς, ο κ. Δοντά μας είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε νέους σχεδιασμούς και προγραμματισμούς. Δεδομένης δε της κατάστασης στον χώρο του γάλακτος θα πρέπει και αυτή την, ε, αυτό το τομέα να εξετάσουμε. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ποιε είναι οι συνθήκε που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί σε πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τεράστιε απώλειε εισοδήματο. Πρέπει αυτή η πραγματικότητα να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, για το δεύτερο πυλώνα είναι πολύ σημαντικό το ότι ενισχύεται με τι προτάσει. Είναι, πιστεύω, εσφαλμένο το να υποστηριχθεί αυτή η επιλογή της εξαγοράς όπως ονομάζεται για τους ελέγχους, ναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον ανταγωνισμό, όλα τα κράτη-μέλη, όλοι οι γεωργοί ουσιαστικά στα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντικό να πληρούνται οι προϋποθέσεις και για να πληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να επαληθεύεται και η πλήρωσή τους. Χρειάζεται λοιπόν ουσιαστικό έλεγχος αλλά όχι στρέβλωση λόγω της γραφειοκρατίας του ανταγωνισμού. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που κάνουν τις προσπάθειές τους να βρίσκονται σε δυσμενές θέσει εναντί εκείνων οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε και μόνο υποφελούνται. Ε, πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει με όσα υπόθηκαν να περάσουμε γρήγορα σε μια απόφαση για την αναθεώρηση κοινή πολιτικής πολιτική. Δυστυχώ δεν βλέπω δεδομένων των προβλημάτων στην, ε, στο πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και δυστυχώ βλέπω ω εκπρόσωπο κράτου μέλου θα έχουμε το περιθώριο να είμαστε έτοιμοι και στο χώρο τη γεωργία μέχρι την επόμενη ε, περίοδο εκμετάλλευσης ε, δυστυχώς. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια παραπάνω. Ευχαριστώ przyjęcia budżetu prosiłbym, aby Pani też rozmawiała z Panią kanclerz Merkel. Για τον προπολογισμό νομίζω ότι θα έπρεπε να το συζητήσετε με την κυρία Μέρκελ καλύτερα. Τώρα ο κύριος Βούς έχει το λόγο. Παόλο Ρούσο. Ιταλικό Κοινοβούλιο. Przepraszamy. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ένα ερώτημα που ήδη έχω υποβάλει και άλλες φορές και που αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά ακόμη περισσότερο αφορά το πρότυπο, το μοντέλο της Ευρώπης που θέλουμε να οικοδομήσουμε και που οικοδομούμε. Ε, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο σε κάτι που επανειλημμένως έχει πει το κοινοβούλιο μας. Θέλουμε δηλαδή την Ευρώπη των ίσων ευκαιριών ή θέλουμε μια Ευρώπη που θα χάσει την ιδιαιτερότητά της και την ιστορία της παραγωγής της. Βεβαίως κατανοώ την ε, διάσταση των επιφανειών ως αξία. Αλλά εάν αυτό δεν συνδέεται και με το εμπορικό ΑΕΠ, τη δυνατότητα να γίνει διαφορά και ισορροπία ανάμεσα στην εξυγχρονισμό και την ε, παράδοση, τη δυνατότητα να ε, επιχειρεί κανείς ε, αλλά ταυτόχρονα να ανοίγει αγορές, τελικά φτάνουμε σε κάποιες άβουλες στάσεις χωρίς να υπάρχει απαραίτητη και έπειτα με συγχωρείτε αν τονίζω το περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Φυσικά είναι πρωταγωνιστής της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά και πάλι τον αποκλείονται οι παραδοσιακές καλλιέργειες της χώρας μας, όπως ας πούμε οι ελαιώνες ή τα κλίματα, ε, νομίζω θα ήταν ε, σφάλμα. Αυτά σχηματίζουν ε, τοπία εδώ και χρόνια. Ίσως να μην είναι σφάλμα, ίσως είναι αδυναμία ανάγνωσης μιας σπουδαίας υπήρου, διαφορετικής από το, το λογικό επίπεδο, από ιστορικό, από γεωγραφικό, χωροταξικό επίπεδο, διαφορετικής από την άποψη την πολιτιστική και την άποψη της νοτροπίας. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση μια κοινή γεωργική η πολιτική, η οποία όμως να πλήττεται από μια κρίση διακυβέρνησης, μια οποιαδήποτε ΚΑΠ, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα έναν μοχλό για εντάσει για αντιρρήσει κατά μια απομάκρης πολιτικής και θα τροφοδοτούσε τον ευρωσκεπτικισμό. Αντιθέτως, χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική που θα αξιοποιεί τι διάφορε ε, ε στην Ευρώπη, θα τονίζει και θα προωθεί την αριστεία, χωρίς να ε, τιμωρεί τις, εκατο... τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που χρειάστηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια να επενδύσουν, να βελτιωθούν, ώστε να εγγυηθούν την ποιότητα των προϊόντων, εγγυόμενη μια απόλυτη ε, ανιχνευσιμότητα. Σας ευχαριστώ. Ο Λόρτ Κανόν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι εγώ ίδιος είμαι αγρότης και το λέω αυτό για να ξέρετε περί τίνος ομιλώ και ελπίζω να δεχτείτε παρόλα αυτά τα σχόλιά μου. Λοιπόν, αν πολλά χρήματα πηγαίνουν από το φορολογούμενο στους γεωργούς, τότε θα πρέπει να υπάρχει και μια αιρεσιμότητα, δηλαδή να ε, υπάρχει προστασία του περιβάλλοντας και να ανταποκρίνεται σε κάποια κριτήρια. Πολλά από αυτά τα ανέφερε ο George Λάιον. Θα ήταν άδικο επίση αν το γεγονό ότι κατά το παρελθόν ένα αγρότη έχει βάλει κομμάτι τη γης του σε περιβαλλοντικό ε, πρόγραμμα να μην μπορεί να υποφεληθεί και να πρέπει να ισχύσει και γι' αυτόν το ίδιο ποσοστό για το πρασίνισμα. Εμείς πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τότε θα πρέπει σιγά σιγά να βάλουμε περισσότερα χρήματα στον πυλώνα 2 αντί για τον πυλώνα 1. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες, πιο μειονεκτικέ, οι οποίες χρειάζονται μια πλήρη στήριξη από εμά, αλλά πρέπει να βάλουμε περισσότερα χρήματα, τουλάχιστον τώρα τον 21ο αιώνα, στην ευρύτερη ύπεθρο, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τις αγροτικές οικογένειε και δεν θα πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε τα προβλήματα που είχαμε κατά το παρελθόν. Χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία, περισσότερη διαφοροποίηση, περισσότερες εκμεταλλεύσεις μικρέ και περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος. Πράγματα που μπορούν κάλλιστα να γίνουν με έναν καλά χρηματοδοτούμενο δεύτερο πυλώνα που πρέπει να αποτελέσει ένα καλό οικονομικό μέσο. Η Επιτροπή μου όμως πιστεύει επίσης, και αυτό δεν το έχουμε πει μέχρι σήμερα, ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους αγρότες από τις θεομηνίες, από τις τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές. Στην Αφρική έχουν ασφαλιστικά προγράμματα με ένα 5% του κόστους για σπόρους ε, ε και άλλα ε, πράγματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί τα προγράμματα αυτά τα ασφαλιστικά είναι πολύ δημοφιλή στην Αφρική. Ελπίζουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει αντίστοιχα προγράμματα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ρόντουστα, έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας ε, παρακαλούσα πάντως ε, να τηρείτε και τη σειρά των τοποθετήσεων όπως έχουν ζητηθεί και να μην είστε αφαίρετο στι επιλογέ σα, γιατί έχω ζητήσει το λόγο από την αρχή αρχή της συζήτησης και μόλι τώρα μου τον δίνετε. Όχι και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Πολλές φορέ το έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως τώρα περάσουμε στην ουσία. Έχει κάνει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε να την εξετάσουμε και το ότι γίνεται αυτή η πρόταση, το ότι έχουμε να την εξετάσουμε οφείλεται στο γεγονό ότι η κοινωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία μάλλον δεν ακολουθεί απαραίτητα τι σκέψει προτάσεις και ιδέες της Γεωργικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μας ζητεί να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό να έχουμε το 30% των άμεσων πληρωμών για την ε, οικολογικότερη παραγωγή, ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφοροποίηση στις παραγωγές, ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, προτεραιότητα στις σχετικές εκτάσεις, στις εκτάσεις δηλαδή με διαφοροποιημένες καλλιέργειες. Πώς θα γίνει όμως αυτό. Εγώ θα προτείνω συναδέλφους να μην νομίζουν ότι είναι κάτι το απλό αυτό ή ότι είναι εύκολο να περάσει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα όριζε ότι διατίθεται τα 58 δισεκατομμύρια που χρειάζεται η Γεωργία. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη προεξαγγείλει περικοπές στο γεωργικό προϋπολογισμό. Γενικότερα περικοπές στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σας διαβεβαιώ ότι πρώτα, θα, πρώτα θύματα θα πέσουν στις περικοπές αυτές ο γεωργικός προπολογισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη πέθρου και τα διευθυντικά ταμεία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σαφείς και να φροντίσουμε ε, να διατυπώσουμε ξεκάθαρα την απέτηση ότι θέλουμε και καθαρά και υγιή, και καθαρό και υγιές περιβάλλον. Για το κάπιν, για, τις τα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις, ήδη έχουν ε, γίνει ψηφοφορίες και στην Επιτροπή Γεωργίας και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ψηφοφορίες οποίες είχαν αποτέλεσμα να βγει από την ε, ε, να, να βγει από τον προγραμματισμό της γεωργικής πολιτικής το ε, κάπινγκ, το, το επίπεδο δηλαδή για τις ενισχύσεις και ότι το 75% των συναδέλφων βουλευτών έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κάπινγκ και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εγκριθούν οι προτάσεις του κυρίου Κάπουλα Σάντος. Είναι μια ευκαιρία, δεν πρέπει να τις ε, απορρίπτουμε. Δεν θα καταφέρουμε διαφορετικά να περάσουμε σε ουσιαστικά μέτρα. Για την κατάργηση της ε, γραφειοκρατίας που ζητήθηκε εδώ, ναι, χρειαζόμαστε βέβαια την, ε, αυτόν τον έλεγχο τη ουσιαστική στήριξη των προποθέσεων, αλλά δεν θέλουμε και τον έλεγχο του, ελέγχο, του ελέγχοντο. Και γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κοιτάξουν από πλευρά του αν μπορεί να διατυπωθεί κατά διαφορετικό τρόπο ο έλεγχο, ώστε να μην ε, όταν ε, είναι υπερβολική η έλεγχη. Νομίζω ότι οι προσπάθειές μας μπορούν να διώσουν ένα πολύ καλύτερο ε, πρόγραμμα για την αναθεώρηση κοινωνικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος, με συγχωρείτε, αλλά με την αλλαγή της, ε, του Προεδρεύοντος εδώ στο Προεδρείο ε, έγινε αυτό το μπέρδεμα. Θέλησαμε να δώσουμε και μια προτεραιότητα στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Γιούργκελ από την, Γιούργελ από την ε, ε, Πολωνική Βουλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συστήσουμε εδώ το μέλλον ε, της γερουκής πολιτικής. Εμείς συζητήσαμε και τελευταία φορά τον Οκτώβριο από πλευράς της Πολωνικής Βουλής. Και πιστεύουμε ότι η απουσία λύσεων η ομοιόμορφη ε, διατύπωση των ε, λύσεων για τις άμεσες πληρωμές είναι μια πολύ κακή επιλογή. Ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι δεν υπάρχει απλούστευση, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην κατανομή των αμέσων πληρωμών και έτσι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση ορισμένα κράτη-μέλη. Τα δε ποσά κατανέμονται όχι με αντικειμενικά κριτήρια, κοινά για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά με βάση ιστορικά λεγόμενα κριτήρια. Βάσει δηλαδή των ε, δεδομένων του παρελθόντος και των πόρων που έχει εισπράξει κάποιο κράτος στο παρελθόν. Ε, η Επιτροπή ε, μιλάει για κάποια διόρθωση προς τις ανισότητες, παρόλα αυτά παραμένει στο κριτήριο το ιστορικό ως βάση των υπολογισμών της, πράγμα το οποίο βρίσκουμε, κρίνουμε ως μια άδικη μεταχείριση. Χρειάζεται μια ισότιμη αντιμετώπιση των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη περιλαμβανομένη και τη Πολωνία που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίε. Και το να παραμένει άδικο και άνισα κατανεμημένο το σύστημα αυτό, που άλλωστε επισήμαναν και οι Πολωνοί συνάδελφοι πριν από μένα, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, ε, αντιβαίνει στην αρχή της ε, αποφυγής των διακρίσεων εις βάρος των γεωργών. Άρθρο 18 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον δε αντιβαίνει στο άρθρο 48 της Συνθήκης. Επίσης μπορούν να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των γεωργικών και περιφερειακών και ε, των γεωργικών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου μέσα στο ίδιο κράτος μέλος και όχι μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει ωστόσο να προβλέψουμε μια λύση που να μην οδηγεί σε άνηση αντιμετώπιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εμείς περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εστερνίσει το στόχο της ισότιμης μεταχείρισης των γεωργών. Τελευταία παρατήρηση, το Πολωνικό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις ποσοστώσεις για το γάλα η κατάργησή τους θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση ορισμένων εκμεταλλεύσεων. Το ίδιο για την ποσόστοση στη ζάχαρη, η οποία πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να αυξηθεί. Μέχρι τα 17 εκατομμύρια τόνων, ποσού το οποίο μας επιτρέπει να διατηρήσουμε αυτάρκεια στην προμήθεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει υιοθετηθεί σωστή λύση προ τη ζάχαρη από το Ευρωπαϊκό. Πρόεδρος διακόπτη. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα ήθελα να συνεχίσω λίγο ακόμα. Μια φράση μόνο. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρέπει και εδώ να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Οι ισχύουσες λύσεις δεν εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία των, των συστημάτων. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Αν ο καθένα μιλάει το διπλό από το χρόνο που έχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν όλοι το λόγο. 1,5 λεπτό από εδώ και πέρα ο καθένα. Ο εκπρόσωπο του Ισπανικού Κοινοβουλίου, ο κύριο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για έναν τομέα στρατηγική σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την γεωργία λοιπόν που διασφαλίζει επισητιστική αυτάρκεια, διασφαλίζει γενικότερα ασφάλεια και επιτρέπει και στον κόσμο να παραμένει στην Ήπεθρο. Εγώ έρχομαι από ένα χωριό πάρα πολύ μικρό και είμαστε οι πρώτοι που ενδιαφερόμαστε να κρατηθεί ο κόσμος στη γη του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί ο προπολογισμό για την γραμμή αυτή. Και είναι τόσο σημαντικό μάλιστα επειδή δεν χρησιμοποιείται το 30% για το πρασίνισμα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί το περιβάλλον, αλλά από την άλλη μεριά να μην επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο με το κόστος οι γεωργοί ή να μην μπορέσουν να έχουν ε, τα εισοδήματα που τους αξίζει βάσει της δουλειάς που προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τώρα να έρθω λιγάκι στο θέμα της ενσωμάτωσης των νέων γεωργών στην ε, δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ε, σήμερα. Για μας είναι πολύ σημαντικό οι γεωργικές αγορές να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στις επαγγελματικέ οργανώσεις των γεωργών και τα μέτρα να είναι πιο αποτελεσματικά. Εμείς θέλουμε επίσης να μειωθεί η γραφειοκρατία όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ. Ναι, φαντάζομαι ότι εμένα εννοείται. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να επικεντρωθώ σε μερικά σημεία που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, λέει εκπρόσωπος ε, του Βελγίου Βαλονία. Πρέπει μεσοπρόθεσμα να περιορίσουμε τα μέτρα ρύθμισης όπως είναι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και να ξαναδούμε και τους διεθνείς κανόνες οι οποίες καθορίζουν τη δικιά μας γεωργική πολιτική. Αντί για τους κανόνες του ΠΟΕ που μιλάνε για τις εξαγωγές πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο την επισητιστική κυριαρχία η Επιτροπή προτείνει διάφορους μηχανισμούς και πρέπει να συνεχίσει να προτείνει μηχανισμούς διαχείρισης με συγκεκριμένα όμως μέτρα που να έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες για να μπορέσουμε όλοι να υποφεληθούμε από τις προσπάθειες που κάνουν για να καλύψουν την ε, ζήτηση με τη δικιά τους προσφορά. Εγκάρσια πρέπει να δούμε τα μέτρα. Η διεύθυνση πάντως που παίρνει η Επιτροπή με το Πρασίνισμα είναι θετική, παρόλο που δεν γίνεται το ποιοτικό άλμα που θα έπρεπε. Παραμένουμε σε, μια, σε ένα σκεπτικό ε, καλών πρακτικών προς την κατεύθυνση αυτή. Έπειτα οι πληρωμές με τα τρία περιβαλλοντικά κριτήρια ε, δεν μας ικανοποιούν. Θα πρέπει όλες οι πληρωμές να έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα και να καθορίζονται και εθνικά και περιφερειακά και όχι να επιβάλλουμε ε, εκ των άνω ε, μέτρα τα ίδια για όλους. Το θέμα της κατανομής των πόρων πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο, βάσει των προσπαθειών που κάνουν οι αγρότες. Θα μπορούσε να υπάρχει μια βασική ενίσχυση στο εισόδημα που να λαμβάνει υπόψη την δουλειά του αγρότη και από την άλλη μεριά να υπάρχει και ένα ποσοστό περιβαλλοντικό που να καθορίζεται βάσει κυπωνικών αρχών κτλ. Οι αγρότες έτσι κι αλλιώς είναι στην καρδιά του ζητήματος έπειτα να μπορούμε να παρεύουμε με μια ειδική στήριξη στους αγρότες, εκείνους που έχουν μια βιολογική παραγωγή, που βοηθούν να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά κλπ. κλπ. Τέλος, και δεν είναι και καινούριο, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να βάλει νέε βάσει για τη σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή και τον παραγωγό. Δεν θα βαθύνω περισσότερο, αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται στι μελλοντικέ πρόπτικε και πρέπει να τολμάει περισσότερο και να μην παραμείνει σε δράνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Στιούαρτ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο, αντίθετα από του περισσότερου συναδέλφου εδώ. Σύντομα για το πρασίνισμα. Αυτέ οι οικολογικέ ζώνε εγώ έχω μια υποσημείωση του, μάλλον μια παράθεση του Επιτρόπου Τσόλο που λέει ότι θα περιλάμβανε τη γη σε περιβαλλοντικό προγράμματα. Ναι, λένε κόσμο, τα έχουμε δει το τις ταινίε, αλλά πρέπει να δούμε και το σχετική νομοθεσία. Τώρα όσον αφορά την διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν είναι πράσινο το να αυξάνεται η αρρώσιμη γη στου δρόμου, ούτε είναι πράσινο οι αποθηκευτικοί χώροι που χρειάζονται επηρεάζονται για τι καλλιέργειε. όλα αυτά θα επηρεάσουν τόσο τι μικρέ, όσο και τι μεγάλε εκμεταλλεύσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν τα θέλουμε αυτά στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν δεχόμαστε την ε, αρρώσιμη μονοκαλλιέργεια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όσοι έχουν ε, και άλλου είδους καλλιέργειες όπως ας πούμε πτυνοτροφία θα πρέπει να θεωρείται αυτό ως διαφοροποίηση της καλλιέργειας. Ε, έγινε και μια πρόταση για πρωτεϊνικές καλλιέργειες. Δεν με εντυπωσιάζει όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σπόρων, ωστόσο θεωρούνται, θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωτικά μια κακή ιδέα, αλλά μπορεί να είναι πρόκληση για τον ένα λεπτό και 41 δευτερόλεπτα. Οι υπόλοιποι σημειώστε το. Σα ευχαριστώ πολύ. Μάκιντάιρ. Μάκιντάιρ ε, είπατε, εννοούσατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ στα προτινόμενα μέτρα πρασινίσματο τη Κομισιόν και τι επιπτώσει του. Εγώ καλωσορίζω τα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου εδώ σήμερα και τι συμβολέ του. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύεται εδώ από, το, από εξαίρετου συναδέλφου από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και έχουν κάνει πολύ χρήσιμε εκθέσει και τα δύο σώματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία UNICEF λύση για τα περιβαλλοντικά μέτρα. Εγώ πιστεύω πως η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να μπορέσουν να φτιάξουν τέτοιου είδους περιβαλλοντικά προγράμματα ώστε να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες πραγματικότητες. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υπάρχει στον Ε.Β. είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη και ήδη είδαμε να βλάπτονται αυτά τα προγράμματα γιατί οι γεωργοί προέβλεψαν τα μέτρα πρασινίσματα που αυτή τη στιγμή προτείνονται. Τα μέτρο πολυκαλλιέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που έχει στόχο. ενδιαφέρον δεν διάβασα τις εκθέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και βρίσκω πως οι χώρες που είναι τόσο διαφορετικές όπως η Φιλανδία και η Ιταλία να συμφωνούν πως αυτό το πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει. Πολύ συχνά εδώ βλέπουμε τις επιπτώσεις του νόμου των παράπλευρων πολιών δηλαδή και των μη ε, ηθελημένων συνεπειών αύξηση της γραφειοκρατίας και κόστους αυτής και διατήρηση, μάλλον και κατάργηση κάποιων εξαιρετικών υφιστάμενων προγραμμάτων. Θα μειωθεί η παραγωγή τη στιγμή που όλοι ανησυχούμε για την ασφάλεια στα τρόφιμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Λίντερμαν. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, τα κρατήδια τη Γερμανία παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή τη μεταρρύθμιση τη κοινωνική πολιτική και θέλουν να τη διαμορφώσουν. Στη Γερμανία τα κρατήδια είναι εκείνα τα οποία ε, λαμβάνουν τι αποφάσει για την υλοποίηση και που αισθάνονται βέβαια και άμεσα τι συνέπειε από την εφαρμογή της ε, συμφωνίες. Βλέπω μεγάλες διαφορές, αποκλείς απόψεων ε, ως προς την προσέγγιση στην κοινή γεωργική πολιτική. Χρειάζεται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για τη γεωργία και την υπεθρό της Ευρώπης, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε πρόκληση, κάθε νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει δεκτή. Πρέπει η πρόκληση μεγάλη των, της πανίδος των ε, φυσικών πόρων να ε, αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και χρειαζόμαστε για το μέλλον μια γεωργία υπεύθυνη, μια γεωργία παραγωγική, μια γεωργία η οποία με υπεύθυνο τρόπο θα αντιμετωπίσει τους φυσικούς μας πόρους. Και σε αυτό, εν συντομία, θα έλεγα μέχρι που μπορούμε να πάμε προς την οικολογικότερη παραγωγή, το greening, δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε επιπλέον περιορισμούς και ρυθμίσεις στη γεωργική πολιτική και μάλιστα να συνοδέψουμε αυτού του περιορισμού και τι ρυθμίσει με άμεσε πληρωμέ, επιδεινώνοντα ακόμη περισσότερο το γραφειοκρατικό φόρτο για του ε, για τους παραγωγούς το 7% που ορίζεται για, τη γεωρική, για τις γεωρικές επιφάνειες θα όχι σαν αποτέλεσμα σε σύνολο Γερμανίας ολόκληρη η, η ολόκληρο το Βίτερμπουργκ να βγει από την γεωργική παραγωγή, να καταλήψει την γεωργική παραγωγή. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε είτε πρόκειται για, τον, για τα πρωτεϊνούχα, είτε πρόκειται για τις εκτατικές καλλιέργειες, μια διαφορετική λύση. Χρειάζονται μέτρα τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ε, ε, για την γεωργική παραγωγή να, αντι... να τροποποιηθούν ώστε να φέρουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα και, κυρίε και κύριοι, καταργήθηκε πριν από μερικά χρόνια η υποχρεωτική αγρανάπαυση για κάποιους λόγους και ήταν σωστή η κατάργηση αυτή. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να εισαγάγουμε τέτοια μέτρα και πάλι στην γεωργική μας πολιτική. Θα έχουν μόνο αντιπαραγωγική ενέργεια. Ευχαριστούμε. Ναι, κυρία Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ την ευκαιρία που μου δίνετε να συμβάλλω σήμερα και σας ευχαριστώ για αυτήν. Είναι σημαντικό κατά τη συζήτηση τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική να τονίσουμε τη στήριξη για την γεωργική βιομηχανία και να διευκολύνουμε την στήριξη στην παραγωγή καθώ και μέτρα τα οποία δεν μειώνουν, ή ε, δεν ε, θα του κίνδυνο την ε, βιομηχανία τη γεωργία ούτε και την βιομηχανία τροφίμων. Εγώ αντιπροσωπεύω μια περιφέρεια τη Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι σημαντικό η απλοποίηση των κανόνων και των κανονισμών για το σύστημα πληρωμών γιατί αυτή τη στιγμή στιγμή για την ε, ενιαία πληρωμή είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα με πολλές επιθεωρήσεις και οι πληρωμές για το 2011 δεν έχουν ακόμα γίνει. Το σύστημα που θα εγκριθεί επίσης θα πρέπει να, προ... να παρέχει, ε, να είναι αποδοτικό και να δίνει την έμφαση στον ενεργό αγρότη, ιδιαίτερα εκεί όπου πολύ ε, γη Ε, είναι αντικείμενο εκμίστοσης. Θα πρέπει λοιπόν η καινή γεωργική πολιτική να μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίμη. Από τη Σουηδία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο όσα είπε η κυρία Όσκαρσον, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε για όλους. Υπάρχει και ο σε ένα να βρεθεί σε ε, σύγκρουση με τον πυλώνα 2. Το πρασίνισμα προβλέπεται στον πρώτο πυλώνα. Έτσι λοιπόν 30% για την ε, πιο οικολογική παραγωγή ως ποσοστό μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Μπορεί από την άλλη να οδηγήσει, σε συνέπεια, σε σημαντικές, ε, σημαντικά ωφέλη για ορισμένα κράτη-μέλη, όταν αυτά είναι καλά προετοιμασμένα, όταν έχουν ε, όμως πολλές ελλείψεις μπορεί να χάσουν σημαντικά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε την γραφειοκρατία και όταν πρόκειται για μεταφορά κονδύλιων από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1 μπορούσαμε να προβλέψουμε άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά ε, για τα κράτη που θα ήθελαν να συνδυάσουν τον, ε, την υποστήριξη. Όμως αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι μια καλή λύση για το μέλλον. Πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση ε, να, επιλέγουν αν θέλουν να γίνει μεταφορά των κονδυλίων και όχι να γίνεται αυτή αυτόματα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Κάτινμπαχ. Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι σήμερα το λόγο τον δίνεται όποιος, ε, ο, ο, τελευταίος έρχεται πρώτος. Έτσι λοιπόν και ο πρώτος τελευταίος βέβαια. Ε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες. Εγώ είμαι σκιώδης, ήμουν συγητής σκιώδης για ε, ε, για την οικολογική διάσταση, για την Επιτροπή Υγείας και Δικαιωμάτων του Καταναλωτή για την ανάπτυξη της Υπέθρου. Ε, ακούω τους συναδέλφους που εκφράζουν τα εθνικά τους κοινοβούλια. Εγώ προσωπικώς θέλω να υπογραμμίσω τα εξή τρία. Πιστεύω καταρχάς ότι χρειάζεται το 30% των μέτρων ε, της οικολογικότερης παραγωγής στον πρώτο πυλώνα, όχι μόνο γιατί θέλουμε και χρειαζόμαστε τη βιοπικιλότητα, όχι γιατί τη χρειαζόμαστε για να ανατρέψουμε σε ένα βαθμό τι συνέπειε των ε, κλιματολογικών αλλαγών, όχι μόνο γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020, αλλά και για να είναι πιο αποδεκτή η χρήση των ε, κονδυλίων, δηλαδή των χρημάτων του φορολογούμενου από την ευρύτερη κοινή γνώμη. Δεν πρέπει να λησμονούμε, δηλαδή όταν συζητούμε όλα τα θέματα αυτά, το μέλλον που θα έχουν οι γεωργικοί προπολογισμοί. Το 7% για, τις, ε, για την οικολογική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η διαφοροποίηση στις καλλιέργειες. Στο δεύτερο πυλώνα επίσης πρέπει το 30% ίσως και 35 ακόμα, δηλαδή αύξηση των κονδυλίων για τα περιβαλλοντικά μέτρα να εισαχθεί και νομίζω ότι η ασφάλιση κινδύνου θα πρέπει να πάει στον πρώτο πλήρωμα και στο δεύτερο. Για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ήθελα να παρακαλέσω να αναλογιστούν το πώς διατέθηκαν ή εάν διατέθηκαν σωστά τα χρήματα στο προηγούμενο διάστημα, στα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της, ε, παραγω... της γεωργικής παραγωγής, της γεωργίας μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερα κονδύλια πώς έχει διάθεσή τη. Έτσι λοιπόν και εν ώψη διάφορων περικοπών που προεξαγγέλλονται, δεδομένου ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να διαθέσουν προπολογισμό αντίστοιχο με τις ε, ε, φιλοδοξίες μας για τη γεωργική παραγωγή θα πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική και ε, πιο ισότιμη κατανομή των κονδυλίων αυτών και τα κράτη τα οποία είναι καθαροί χορηγοί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια στον ε, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για αυτά σχέδια τα οποία υλοποιούνται και αποβαίνουν προ προς των κρατών αυτών. Και επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει και η διάσταση που θα πρέπει να εξετάσουμε με τον φόρο των στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τις τάσεις που είχαν τηρήσει εκεί τα κράτη-μέλη. Δηλαδή χρήματα τα οποία δεν έχουμε δεν μπορούμε να τα αναδιανύμουμε παρά μόνο κατά τρόπο ισότιμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω μόνο ότι ούτως ή άλλως ε, η διοικητική υπηρεσία της Επιτροπής Γεωργίας είναι αυτή που μου έδινε τα χαρτάκια ε, για να δώσω το λόγο στους διάφορους ομιλητές. Και τώρα ο εκπρόσωπος του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Λάπα. Ο κύριος... Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ μια που πιέζει ο χρόνος, εγώ θα επικεντρωθώ πολύ γρήγορα σε κάποια σημεία που με απασχολούν εμένα προσωπικά και που δεν έχουμε συζητήσει αρκετά. Αγροτικές αγορές. Ο εισηγητής είπε ότι πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία της διατροφικής αλυσίδας. Όμως στην Ευρώπη ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί. Γιατί στην διανομή υπάρχουν ε, συμφέροντα και Πιστεύουμε ότι αυτό που προτείνεται εδώ είναι το ελάχιστο και θα έπρεπε να προτείνονται περισσότερα πράγματα. Επίσης, για τη χώρα μας, εμείς θέλουμε να διατηρηθεί ο περιορισμός για ορισμένα προϊόντα, όπως είναι γάλα, ζάχαρη, όμως πρέπει να κρατήσουν τις ποσοστώσεις τους. Θέλουμε επίσης ένα δίκτυο ασφάλειας και μια μέση παρέμβαση για την αποθήκευση και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις και να μην περιμένουμε πρώτα να βουλιάξουν οι γεωργοί. Μεταρρύθμιση ναι, αλλά τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία εισάγουμε από το εξωτερικό τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που επιβάλλουμε εμείς στα δικά μας, θα έπρεπε να υπάρχει αμοιβαιότητα εδώ. Τέλος, η ενεργός γεωργία φυσικά και είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εκείνους οι οποίοι έχουν αυτή τη δραστηριότητα αλλά και την εμπορική. Έπειτα για το θέμα της επιφάνειας αναφοράς, αυτό πρέπει να μπορεί να το αποφασίσει ο καθένας. Τέλος, να περιορίζεται η σύγκληση. Όσον αφορά το πρασίνισμα, πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό και τέλος για τα οικονομικά όρια. Το μοντέλο άμεσων πληρωμών πρέπει να περιλαμβάνει μέσα τα οποία να επιτρέπουν να μην υπάρχουν ε, προβλήματα με τον ε, προπολογισμό, τα χρήματα δηλαδή, τα οποία ορισμένες χώρες μπορεί να θέλουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλεμπά, ε, Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διάκριση όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες των νέων χωρών μελών. Και έχω να ρωτήσω το εξής. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίσει σαφή και με διαφάνεια κριτήρια για όλους τους ε, Ευρωπαίους αγρότες, πότε θα το κάνει, ερώτηση είναι αυτή. Γιατί αλλιώς το μόνο που κάνουμε είναι να διατηρούμε τη διάκριση αυτή. Δεν επιδεικνύουμε αλληλεγγύη, δεν υπάρχει επικουρικότητα, δεν υπάρχει ενιαία αγορά τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, στην Πολωνία φτάνουμε στο 100% των μέσων εξόδων ανεκτάριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην πληρωμή είμαστε κάτω από το 80% και δεν υπάρχει και συμφωνία για μια διαφυροποίηση. Κάτι άλλο το οποίο δεν συζητήσαμε σήμερα είναι ότι με τα σχέδια αυτά κανονισμού πολλές αποφάσεις θα είναι τελικά κατεξουσιοδότηση πράξεις στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν θα πρόκειται για ρυθμίσεις που θα έχουν περάσει από διαβούλευση με τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια έτσι όπως θα έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι αρκετά επεξηγματική όπως θα ήταν τα κράτη-μέλη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Το κριτήριο των θαμινιών. Μπορείτε να μου πείτε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και πώς θα ανακτήσουν τις δυνατότητε τους οι αγρότες, γιατί αυτό που λέμε τώρα είναι ανάκριση του 30% της παραγωγής. Είναι λίγο παράδοξο, γιατί γίνεται διάκριση σε βάρος των αγροτών εκείνων οι οποίοι εκτρέφουν ζώα. Θέλω να ξέρω κατά πόσο υπάρχουν πληρωμές οι οποίες να επιτρέπουν να διασφαλίζουμε και για τα ζώα και για τις ε, καλλιέργειες το ίδιο. Έχουμε όλο και περισσότερες απώλειες τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστούμε. Αυστρία. Ο κύριος Γκρούβερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, Ελπίζω οι προτάσεις των βουλευτών να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και να διατυπωθούν κατά τρόπο και πιο φιλόδοξο. Θα υπενθυμίσω την έκθεση DES και Lions αλλά και την Evans του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις οποίες είχαμε πάρα πολύ καλές προτάσεις, τις οποίες πλέον δεν βλέπω. Στην έκθεση Ντέσε παραδείγματι και στην έκθεση Lions είχαμε μία πρόσβαση ε, στην βιολογική καλλιέργεια, προγράμματα και λύσεις οι οποίες δεν βλέπω να επανέρχονται εδώ. Και μια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει για πρώτη φορά τη συναπόφαση στη γεωργική πολιτική, θα έπρεπε πιστεύω να ε, επιδείξει περισσότερη παρησία και περισσότερη φιλοδοξία ως προς τα τη πρόσπιστη διεκδικήση του. Μην ξεχνάμε ότι ο Ευρωπαίο πολίτη περιμένει και ουσιαστική συναπόφαση και αποφασιστική προσέγγιση, μαχητική προσέγγιση στην κοινή γεωργική πολιτική. Για τον γεωργό, δεδομένων των δυσκολίων που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί, αλλά και για τον καταναλωτή της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κοιτάξουμε το μέλλον στις αγορές. Έχουμε 40 εκατομμύρια τόνους εισαγωμένων τροφίμων στην εποχή που μιλάμε. Ένα δε κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η μη γενετικά τροποποιημένη παραγωγή πρωτεϊνούχων στην ε, οικονομία μας. Κάτι το οποίο τουλάχιστον κατά 10% πρέπει να επιδιώξουμε να εξασφαλίσετε στην Ευρώπη για τις αγορές μας, για τις ε, κλιματικές μας συνθήκες, για το περιβάλλον μας. Χρειαζόμαστε επίσης ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσεως για την οικολογία, για την οικολογική παραγωγή και ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε ενώνοντα το επίπεδο Ε, ανώτατο που θα ξεκινάει στα 150.000 ευρώ αλλά στα 35.000 ευρώ για να έχει ουσιαστική λειτουργία αυτή η προσπάθεια. Όπως είπε και ο κύριος Δες, ε, η ενοποίηση των πληρωμών πρέπει να γίνει ταχύτατα. Διαφορετικά θα πρέπει να εξηγήσουμε στον καταναλωτή, στον γεωργό, πράγματα ανεξήγητα. Η γεωργική ανάπτυξη, ανάπτυξη πέθρου είναι επιταγή τη σύγχρονη εποχή και δεν βλέπω ουσιαστική πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Δεν βλέπω ουσιαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόκκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται να τοποθετηθώ και εγώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκή ε, βαθμό φιλοδοξία στις προτάσει αυτέ Είναι περίπλοκες, δεν βοηθούν ούτε το περιβάλλον, ούτε το ανταγωνιστικό, το μακροπρόθεσμα ε, του κλάδου. Δεν αποδίδουν τα κονδύλια που θα διατεθούν και θα οδηγηθούμε τελικά στι σημαντικέ περικοπέ στον προπολογισμό του πρώτου πυλώνα. Και ενώ προτείνεται η κατάργηση κάποιων ε, πυλώνων από τον, κάποιων αξώνων μάλλον του πρώτου πυλώνα ε, παραμένει πολύ περίπλοκος ο γραφειοκρατικός ο μηχανισμός. Οι γεωργικές δαπάνες για την περίοδο 2014-2020 45,6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχει ακόμη βεβαιωθεί, αλλά θεωρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ υψηλό ποσό και η τάση θα πρέπει να είναι μάλλον η μείωση παρά η αύξηση των ε, διατηθεμένων ε, ποσών. Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι στο πολιτιστικό οικονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπεται η αύξηση των ευρωπαϊκών προπολογισμών. Δεν θέλουμε χωριστά προγράμματα που θα συμφωνούνται χωριστά και που θα οδηγούν σε συνολική αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η ομαδών δημοσιονομικές μεταφορές από τα κράτη-μέλη και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με το βιωτικό επίπεδο των κρατών μελών. Ε, και ενώ δεν μπορώ να πω πολλά λόγω της θέσης ε, που κατέχω στη συνεδρίαση αυτήν και των, ε, των θεσμικών της περιορισμών, θα ήθελα να πω ότι μπορεί κάποια κράτη-μέλη να διαφοροποιούνται και δεν μπορούν να αγνοούνται οι θέσεις τους. Ευχαριστώ, ιδιαίτερα τον Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Ο κύριος Ρούμπιξ. Πρόκειται αυτά τα οποία συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Το θέμα της ε, μεταρρύθμισης είναι στην ημερήσια διάταξη εδώ και δύο χρόνια. Ήδη βλέπουμε, διαβλέπουμε μάλλον το σκελετό αυτής της νέας πολιτικής και συμφωνώ με πολλούς ε, μιλητές, δεν χρειάζεται να επαναλάβω πολλά, αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξή. Οι βαλτικές χώρες και κάποιες ακόμα θέλουν να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή για τον άμεσο πληρωμό. Δεν είναι το θέμα της μόνο ελεύθερης αγοράς. Οι ψηφοφόροι στη Λετωνία με ρώτησαν που την περασμένη εβδομάδα να μιλήσω, μου ζήτησαν να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Οι γεωργοί μας ε, δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Ε, για... Φεύγουν λοιπόν από την Ήπεθρο, πουλάνε τη γη τους και αυτή η γεωργική γη αγοράζεται από πλούσιους από την Δυτική Ευρώπη. Εκεί φυτεύουν δέντρα, κάνουν δασοκομεία και εδώ ταυτόχρονα λέμε ότι εμείς χρειαζόμαστε ασφάλεια τροφίμων. Χρειάζεται να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα. Εγώ είμαι ευγνώμων στον κύριο Ντές και στον κύριο Τσόλος για το τι πέτυχαν σε αυτές τις προτάσεις που ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να διανέμονται πιο δίκαια. Η πρόταση αυτή είναι δικαιότερη από την προηγούμενη ωστόσο δεν αρκεί. Ελπίζω ότι η πρόταση θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και ότι όλοι θα λάβουν τουλάχιστον 80% του μέσου όρου. Ε, η σημερινή πρόταση προβλέπει 65% του μέσου όρου. Παρακαλώ, βρείτε ένα εκατομμύριο για να βελτιώσετε την πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Κύριε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εμείς σε Εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να συζητήσουμε την βάση που παρουσιάζει τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα Εθνικά Κοινοβούλια των ε, διάφορων χωρών μελών. Υπάρχει ένα θέμα που είναι κοινό σε όλες τις χώρες και κοινό σε όλα τα εδάφη που έχουν να κάνουν με την ΚΑΠ. Και αυτό είναι το θέμα της ε, εγκατάλειψης των εδαφών αυτό από τους Ευρωπαίους πολίτες, η κατάληψη της υπαίθρου δηλαδή. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό και θα έπρεπε να υπάρξουν νέα κονδύλια. Και δεν λέω νέα κονδύλια από το δεύτερο πυλώνα, αλλά να αρχίσουμε με την ευκαιρία αυτή να ζητάμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν σε μια νέα διατύπωση. Διατύπωση που έχει να κάνει με όλες μας τις χώρες. Στόχος είναι λοιπόν η διατήρηση του κόσμου στη γη του. Να έχουν δουλειά. Αλλά να βρούμε και εναλλακτικές λύσεις για απασχόληση. Μιλάμε για κονδύλια που δίνονται, αλλά όλο και λιγότερους αγρότες έχουμε στην Ήπεθρο. Και υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε εμείς που είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Μιλάμε μεταξύ άλλων, για δράσεις στήριξης των μικρών δήμων, των μικρών επιχειρήσεων που προσφέρουν απασχόληση κυρίως στις γυναίκες. Μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές και πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στήριξη της απασχόλησης μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Κλείσαμε τον κατάλογο και τώρα οι εισηγητές θα πάρουν και πάλι το λόγο για δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Καπούλα Σάντος. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ γέμισα το σημειωματάριό μου με τις 44 παρεμβάσεις που άκουσα με όλη μου την προσοχή και που ε, αντικατοπτρίζουν τις, σημειώσει που αντικατοπτρίζουν τη συζήτηση που έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα της κατανομής των ενισχύσεων, το θέμα της απλοποίησης της γραφειοκρατίας ήταν ε, τα, τα θέματα που επαναλήφθηκαν ε, Πολάκης, το greening, ευρύτερος ε, κατάλογος, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Όλες αυτές οι ανησυχίες είναι ανησυχίε ανησυχίες που έχουμε και εμείς εδώ συζητήσει ε, εις βάθος. Εγώ προσπάθησα στις εκθέσεις μου να συνο να, να συνθέσω όλες αυτές τις ανησυχίες, ε, να βρω και ένα σημείο συνένεση. Ε, αλλά είναι προφανέ ότι είμαστε ακόμα πολύ ε, μακριά από αυτή την συνένεση που θα χρειαστεί καταρχήν να βρούμε εδώ στο Κοινοβούλιο και έπειτα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωργίας. Όπω θα καταλάβατε, είμαστε όλοι μα βουλευτέ. και σε αυτό το νέο πλαίσιο της συναπόφασης είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει μια θέση ισχυρή και υπεύθυνη ένα κοινοβούλιο ενωμένο είναι ένα κοινοβούλιο που είναι πολύ ισχυρό απέναντι στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Ενώ αν είμαστε διχασμένοι, είμαστε αδύναμοι. Δεν θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες να επηρεάσουμε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και δουλέψαμε σε διάφορες πολιτικές ομάδες προς την κατεύθυνση ε, της ε, ανέβρεσης σημείων και συνένεσης και συνεννόησης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γύρω από τα βασικά θέματα τα οποία αναφέρατε. Γι' αυτό και σε δύο λεπτά βέβαια δεν μπορώ να σχολιάσω όλες τις παρεμβάσεις, αλλά να γνωρίζω θετικές ε, παρεμβάσεις, θετικές ε, συμβολές ε, που και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια τακτική επαφή μέσω της νέας τεχνολογίας, γιατί σήμερα έχουμε πρόσβαση στην ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών με διάφορους ε, τρόπους, ε, να εκτιμήσω ε, και τις γραπτές παρεμβάσεις από, πολλές, από πολλά κοινοβούλια και εγώ φυσικά είμαι στη διάθεσή σας ως συζητητής για την ανταλλαγή πληροφοριών και για περαιτέρω επαφές όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις τροπολογίες των Ευρωβουλευτών μέχρι τις 10 Ιουλίου και έπειτα θα έχουμε και τον ε, Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να, φτάσουμε σε να φτιάξουμε στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ένας ε, χρόνος δηλαδή ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και να καλύψουμε τις δικές σας ανησυχίες. Να σας ευχαριστήσω όλη μια φορά για όλες τις συμβολές που βοηθάνε στη βελτίωση της ε, δουλειάς μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ την δυνατότητα να συνεχιστεί η συζήτηση με τους συζητητές μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ε? Κύριος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Όπως είπε και ο Λουίς, αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την συζήτηση που έχουμε και εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημειώνω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση όσον αφορά το θέμα της κοινή οργάνωσης αγορών. Πάρα πολύ υπογραμμίσατε ότι πρέπει να ενισχυθεί η δύναμη των αγροτών, φροντίζοντας βέβαια πάντα να λειτουργεί καλά η αγορά. Αυτή είναι μια βούληση που συμμερίζεται και η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιος από εσά, νομίζω ο Γερμανός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό και είπε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα. Δεν συμφωνώ. Αντίθετα, στους έξι μήνες που δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα, διαπίστωσα ότι οι διάφορες χώρες μας και οι αρχές για τον ανταγωνισμό ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Το ότι υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές μεταξύ μας είναι αυτό που ζημιώνει την αγορά μας και επιτρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών των χωρών μας. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν σε ειδικέ παραγωγές, τον Ίνο, όπου πράγματι προτείνω και εγώ να φέρουμε και πάλι τα δικαιώματα φύτευση, βέβαια με κάποια ημερομηνία, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 76 που μας υποχρεώνει να βάζουμε ημερομηνία. Μην επανέλθω στο όσο είπαμε για τη ζάχαρη, όσο για τα γαλακτοκομικά. Εμείς και με ακούει και αυτό που ήταν εισηγητής για το πακέτο κάλακτος πριν από λίγο καιρό για να με διορθώσει, ε, πρόκειται για ένα πρώτο διάβημα. Σίγουρα πρέπει να συμπληρωθεί έτσι ώστε ο τομέας των γαλακτοκομικών και αφού σταματήσουν οι ποσοστώσεις να μπορέσει να επιβιώσει παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από τη δική μου πλευρά, όπως ε, και οι προηγούμενοι εισηγητές, ε, θέλω να ευχαριστήσω για όλες ε, τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ θεωρώ ότι είναι διάχετη σε πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις ένα, το ένα έντονο αίτημα το Κοινοβούλιο να ασκήσει πλήρως το ρόλο του συνομοθέτη που έχει και να διατυπώσει με τολμηρό τρόπο σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, προτάσει τροποποίηση ή προσαρμογή στην ε, πρόταση μεταρρύθμισης που υπέβαλε η Κομισιόν για την κοινή γεωργική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, επίσης, ε, σε πολλές παρεμβάσει ε, διαφάνει μια εκτίμηση για την προσπάθεια που καταβάλαμε για απλοποίηση Σήμερα είμαστε όλοι πεπισμένοι πως οι γεωργοί θα πρέπει να ασχολούνται όλο ένα και περισσότερο με τη δουλειά τους στους, στους αγρούς και με τις δραστηριότητες πώληση και εξοπίση των προϊόντων τους και να μην ε, σπαταλάν το χρόνο τους ε, συμπληρώνοντας έντυπα και υποβάλλοντας αιτήματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ορισμένες προτάσεις μπορούν φυσικά να γίνουν δεκτές, αλλά με τη δική σας υποστήριξη και με τις δικές σας υποδείξεις νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα και να μειώσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο σε πολλούς, για πολλούς γεωργούς. Μια τελευταία σύσταση αφορά τη συζήτηση που έγινε για το πρασίνισμα, το greening, greening με περιορισμένες κυρώσεις για την πληρωμή του πρασινίσματος ή greening με κυρώσεις που ξεπερνούν και μπορεί και να κυρώσουν τη βασική πληρωμή. Ήδη στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες όπως θα φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι αυτό θα, αυτή θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση, ένα ανοιχτό θέμα μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ ωστόσο για τις ερωτήσεις και θα επανέλθουμε και εγώ και όπως οι υπόλοιποι ε, εισηγητές θα είμαστε στη διάθεσή σα για προτάσει και σχόλια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του ΣΥΠΗΝ από τα Κοινοβούλια. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Πολλές είναι οι προκλήσεις Κυρίως όμως βλέπω το περιβάλλον ως κύριο θέμα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Για τη Βαλτική είναι σημαντική η ρήπανση από την Πολωνία και τη Δανία, αλλά και τη Γερμανία. Το πρόβλημα άλλωστε δεν έχει σημασία από πού πηγάζει. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για τις άμεσες πληρωμές πρέπει να τις συζητήσουμε. Ε, πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που ζήτησαν νέες και πιο φιλόδοξες ε, λύσεις για τις άμεσες πληρωμές. Και πάνω απ' όλα να επαληθεύεται ότι αυτές δεν πηγαίνουν σε ε, στόχους που δεν ήταν οι αρχικοί. Οι γεωργικές εκτάσεις θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι έχουν μια αξία αναλογική ως προς τις χορηγούμενες ε, άμεσες πληρωμές. και η ενίσχυση που θα δίνεται δεν θα πρέπει να θέτει σε δυσμενέστερη θέση ένα γεωργό ο οποίος ενδεχομένως χρειάζεται ένα δάνειο ή έχει εκτεθεί οικονομικά για να αναπτύξει τι δραστηριότητε του. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να, καταρχάς θα πρέπει να διατηρηθούν οι ιστορικέ αναφορέ, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να περάσουμε σε μια πιο καινοτόμο, πιο εφάνταστη λύση για τι άμεσε ενισχύσει για την ε, πράσινη παραγωγή, αλλά και για μια αποτελεσματική οικολογικά παραγωγή για ένα καλό πράσινο περιβάλλον. Πιστεύω ότι όλοι μας θα μπορέσουμε να βρούμε καλές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Η πολιτική συνοχή και δεύτερος πυλώνας με την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Στη συνοχή αναφέρεται και η διάσταση των αστικών κέντρων, αναφέρονται διαφορετικέ προτεραιότητες, αλλά όχι η χρήση της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη πέθρου. Ο δε πρώτος πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η παρέμβαση που δεν συζητείται επαρκώς παρά τις σημαντικές προσπάθειες του κύριου Ντόντα. Παρέμβαση παραδείγματι στα σιτηρά, στον χώρο των σιτηρών. Που έχει συνέπειες και στην αγορά είτε του βόλου είτε του χείριου κρέατος. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε τις προσπαθίες μας πιστεύω. Και για να κλείσω, πρόβλημα αποτελεί επίση και η ανάγκη για τη δημιουργία νέων μέσων υποστήριξη στην ΠΑΚ έγινε λόγος για επιδοτήσει σε επενδύσεις, ε, σε η δάνεια καλύτερα ή δάνεια για επενδύσεις που έχουν ληφθεί. Το έχουμε ξανασυστήσει αυτό, είναι κάτι το οποίο έχουμε δει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ο Γεωργός να έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει σε ποιο βαθμό ε, τον συμφέρει κάποιο δάνειο ε, με τους όρους που θα το χορηγούν οι τράπεζες και εάν μπορεί να ζητήσει ε, τις επιδοτήσεις επιτοκίου. Ε, επίσης εάν ο προπολογισμό σα φαίνεται ισχυρό, δεν πρέπει και να λησμονούμε ταυτόχρονα ότι είμαστε περισσότερα κράτη-μέλη τώρα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση σα ευχαριστώ όλου για τη συμβολή σα στη συζήτηση. Έχουμε διαφορέ βεβαίω μεταξύ μα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ωστόσο συνένεση. Συνένεση γιατί αυτό περιμένει ο Γεωργός, αυτό περιμένει η Ευρώπη. Είμαι βεβαίως ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο δε ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σημαντικά ε, ενισχυθεί. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Καλό όλους τους εδώ σε μια δεξίωση άτυπα, ένα ποτηράκι να πιούμε μαζί, εδώ στην έξοδο, βγαίνοντας από την αίθουσά μας. Ε, θα έχουμε ακόμη μια ευκαιρία για συζήτηση μεταξύ των συντονιστών για 5-10 λεπτά. Γι' αυτό παρακαλώ όσοι δεν είναι συντονιστές να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Και παρακαλώ να παραμένει το προσωπικό όταν όσο χρειάζεται, στο βαθμό που χρειάζεται για την συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις προσπάθειες για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη.